Sí, a ver, vamos a empezar la reunión porque hay personas que tienen. Bueno, les pido por favor que tomen asiento a todos porque vamos a empezar la reunión. Siento levantar. Η συνεδρίαση και συγγνώμη που φωνάζω λίγο είναι μόνος τρόπος να με ακούσετε. Θα αρχίσουμε με το σημείο 14 της ημερησιδέξης ανταλλαγή απόψη με κρουσόπ στο ΜΕΑ επί του θέματος της πειρατείας των Ινδικό ωκεανό. Ε, ε, Όπως γνωρίζετε, καλέσαμε κάποιον εκπρόσωπο της επιχείρησης Αταλάντα. Δυστυχώς ζήτησαν συγγνώμη λέγοντας ότι φέτος, ε, ε, αυτό το μήνα στις 16 θα υπάρχει κοινή ακρόαση μεταξύ των Επιτροπών Αλίας Μεταφορών και Αμυνάς, όπου θα είναι εκεί ο υπεύθυνο ε, της ε, επιχείρησης Αταλάντη. Εστάλει όμως εκ μέρους του Συμβουλίου ένας παρατηρητής. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω, δεν ξέρω από τους παρόντες εδώ ποιος είναι. Εν πάση περιπτώσει η γραμματεία θα το λάβει υπόψη, αν θέλει μπορεί να λάβει το λόγο, επειδή δεν είναι όπως σας είπα ο Δυνάβροχος Με τον κύριο Μπουσόν, εκπρόσωπο της Κονχέλ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της ε, Γαλλικής Ένωσης του Κατευσιμένου Τόνου, επίσης έναν ε, συνάδελφό σας από την ε, Ισπανία καλέσαμε, δεν είναι παρόν. Κύριε Μπουσόν, θα μας παρουσιάσετε τα προβλήματα. Ξέρετε ότι μπορείτε να παρουσιάσετε τις απόψεις όλων και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα πειρατείας και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλοίο, το Αλακράνα, το Ισπανικό, το οποίο έχουν ε, ακινητοποιήσει οι πειρατές από τις 2 Οκτωβρίου. Ο κύριος Καντέκ επίσης, που θα είναι εκπρόσωπος της Επιτροπής μας στην κοινή ακρόαση, μπορεί να μας παρουσιάσει και κάποιες απόψεις του κλάδου σήμερα. Ο κύριος Μπουσόν λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε για να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα της πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό. Έχω κάνει μια μικρή παρουσίαση συνοπτική και να σας πω περί τίνος πρόκειται. Είναι οι διαφάνειες μου αγγλικά, αλλά εγώ θα μιλήσω γαλλικά βεβαίως. Μιλούσατε, κύριε Πρόεδρε, για το Αλακράνα, που είναι το πλοίο που βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια, που προσπαθεί να ξεφύγει από ένα τακίφ που προσπαθούν να προσεγγίσουν. Θα χωρίσω την ομιλία μου σε τέσσερα μέρη. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η κατάσταση σχέση με την πειρατεία. Δεύτερον, ποια είναι τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στον κίνδυνο αυτό της αυξανόμενης πειρατείας. Τρίτο παρατήρηση, συμπληρωματικότητα όλων των μέτρων αντίδρασης και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον. Το τέταρτο μέρος. Το 2008 πρέπει να πω ότι η πειρατεία περιοριζόταν στον κόλπο του Άδεν. Στο τέλος του 2008 επεκτάθηκε και στην περιοχή της Λεκάνης της Σομαλίας. Αρχές σε 2008 το πλάια παγίω, το ισπανικό πλοίο επίσης είχε υποστεί μια προσπάθεια προς τους πειρατές και το Ντομενέκ αργότερα ένα γαλλικό πλοίο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2008 Euh, Αυξήθηκαν οι πειρατές των πειρατών στην περιοχή αυτή της Λεκάνης Σομαλίας και σε σχέση με τον προηγούμενο χάρτη βλέπετε εδώ ότι οι πειρατές έφτασαν και εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των Σεϊχελών και την ξεπέρασαν. Έφτασαν πολύ κοντά λοιπόν στην ακτή της Σομαλίας. Πώς έχει η κατάσταση. Πάρα πολλές επιθέσεις στην περιοχή αυτή των, ε, στις Σεϊχέλες, οι πειρατές. Ποια στρατηγική ακολουθούν. Περιμένουν τα πλοία, τα οποία θα κάνουν σταθμό στο Μάη. Έτσι βλέπετε την εξέλιξη των επιθέσεων πειρατών από τον Αύγουστο του 2008. Έχετε τον συνολικό αριθμό επιθέσεων τις οποίες μπορέσαμε να καταγράψουμε, Ανάλογα με τι πηγέ που έχουμε, οι αριθμοί μπορούν να έχουν κάποια απόκληση. Εδώ εμπνεύστηκα από τι γαλλικέ στρατιωτικέ πηγέ. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία περίοδος ε, των μουσώνων, Ιούλιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, την οποία δεν έχουμε πολλές επιθέσεις πειρατών, αλλά σε σχέση με πέρσι το φθινόπωρο έχουμε πολύ λιγότερες ε, επιθέσεις πειρατών στον κόλπο του Άντεν, αλλά αντιθέτως έχουμε το 2009 αύξηση, όπως σας είπα, στη λεκάνη της Σομαλίας και σήμερα έχουν αντιστραφεί οι αναλογίες μεταξύ ε, λεκάνης της Σομαλίας και κόλπο του Άντεν. Πρέπει επίσης να διευκρινίσω το εκρή. Δεν θα σας κάνω τώρα λεπτομερή εξήγηση των επιπτώσεων για την αλία, ότι πες το Μάρτιο είχαμε πει πόσο ευάλωτα είναι τα πλοία μας. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Τα τρία τέταρτα των αλληλευτικών ζωνών μας σήμερα βρίσκονται στην ε, ζώνη, αυτή που βλέπετε με τις στικτές, ε, δηλαδή εκεί που είναι η περιοχή στην οποία έχει αναπτυχθεί η επιχείρηση Αταλάντη. Εμείς λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτή τη ζώνη με τη διαγράμμιση και η Αταλάντη τι συστήνει να αποφεύγεται αυτή η ζώνη. Τα ψάρια τον περισσότερο καιρό κινούνται εντός αυτής της ζώνης. Ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Στο τέλος του 2008 χρησιμοποίησαμε ένα, ένα αέρια μέσα του ναυτικού της Ισπανίας αισθάνθηκαν πιο μεγαλύτερη ασφάλεια και συνέχισαν αυτή τη δραστηριότητα μετά το τέλος, πως το τέλος του έτους είπαμε. Μετά, λόγω των ε, ψαριών, βγήκαμε λίγο από τις ζώνες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πειρατές. Από το Φεβρουάριο είμαστε στην περιοχή της ζώνης Μοζαμβίκης και μετά αυξήθηκαν οι επιθέσεις των πειρατών, για τις οποίες σας εμίλησα, μετά το Φεβράριο λοιπόν, το δεύτερο τρίμηνο, με πολύ σημαντικό αριθμό επιθέσεων εντός λεκάνης Σομαλίας και εντός της οικονομικής αλλιευτικής ζώνης των ε, Σέιχελών και κοντά στις ακτές της Ταζανίας. Η Αταλάντα βοήθησε, Αταλάντη βοήθησε πολλά πλοία να βγουν εκτός ζώνης υπήρχε και υπέρπτυση αεροπλάνων για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε τα πειρατικά πλοία και τα σκιφ και έγιναν και κάποιες συλλήψεις. Παρ' όλα αυτά, επεκτάθηκαν οι ζώνες επιθέσεων των πειρατών, φοβήθηκαν οι ναυτικοί Και δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε, κανένα εφοπλιστής δεν ήθελε τα πλοία του να δραστηριοποιούνται εκεί, δεδομένου ότι και οι ίδιοι ναυτικοί αρνούνταν σε τέτοιες επικίνδυνες ζώνες. μία από τις πρώτες αντιδράσεις ήταν κάποια πλοία να φύγουν από τον Ινδικό ωκεανό, να πάνε στον Ατλαντικό, στα πλαίσια των ε, διαθεσίμων ε, αδειών που είχαμε για λίευση στον Ατλαντικό και η Γαλλία ζήτησε στην κυβέρνησή της προστασία. Προστασία που μας χορηγήθηκε και από την 1η Ιουλίου του 2009 έχουμε στρατιωτικούς πάνω στα πλοία, πράγμα που επέτρεψε στις αλληλευτικές δραστηριότητες να επαναληφθούν και κυρίως μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης με τους ναυτικούς οι οποίοι λέγουν όταν ερωτώνται ότι και πάλι μπορούμε να αλλιεύσουμε χωρίς να ανησυχούμε για τους πειρατές δεδομένου ότι έχουμε ε, στρατιωτικούς στο πλοίο και θα μας υπερασπίσουν. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Για αλίες και ναυτικοί πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, επαγρυπνούν για να μην πλησιάζουν οι πειρατές, αλλά δεν θέλουν να πάρουν και υπέρμετρους κινδύνους. Από τότε λοιπόν που έχουμε στρατιωτικούς, επτά επιθέσεις έγιναν και πώς τελείωσαν με καταδίωξη των πειρατών. Έγιναν κάποιοι πυροβολισμοί προειδοποιητικοί για να καταλάβουν ότι υπήρχαν στρατιωτικοί έτοιμοι να αναχαιτήσουν την επίθεση, στην ε, αρχή χρησιμοποιήθηκαν ε, κάποιοι ε, βολές φωτεινών σημάτων. Νόμιζαν ότι ήταν κάτι διαφορετικό, ότι ζούσαν βοήθεια οι ευρισκόμενοι στο πλοίο οι πειρατές. Και μετά κατανόησαν ότι ήταν μόνο μία προειδοποίηση. Μπορούσαν να ρίξουν και πραγματικά πύρα. Έτσι λοιπόν φεύγανε κάθε φορά τις τελευταίες φορές οι πειρατές. Εδώ σε αυτή λοιπόν την ε, διαφάνεια σας δίδω, εξηγώ πως έχουν τα πράγματα όσον αφορά τους, ε, τον στόλο, τον αλλιευτικό για τον τόνο. Δεν είναι εδώ οι Ισπανοί συνάδελφοι. Ποιο είναι ο δικό μα στόλος. Δέκα πλοία με στρατιωτικούς και πέντε τα οποία μετέφεραν τη δραστηριότητά του στον Ατλαντικό ωκεανό. Επίσης στην δική μα την οργάνωση έχουμε και ένα Ιταλική σημαία πλοίο το οποίο προσπαθεί να τύχει στρατιωτικής προστασίας. Όσον αφορά τον αλλιευτικό στόλο των Ισπανών, Επιβεβαίωσαμε τους συναδέλφους ότι τα 13 πλοία, τα ισπανικά, σύντομα θα έχουν ε, ιδιωτική ασφάλεια για την προστασία τους. Δεν είναι ο Χωσέ Άγχελ εδώ πέρα, δεδομένου ότι έχει κάποια συνάντηση με τις ε, αρχές τις στρατιωτικές και οι Ισπανοί συνάδελφοι επίσης μετέφεραν κάποιες δραστηριότητες ε, επτά πλοίων στον Ατλαντικό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι επίσης είναι υπεύθυνη τη διαχείριση κάποιων αλλιευτικών πλοίων από τις Σεϊχέλες, εννέα από τα οποία έχουν ε, ιδιωτική φρουρά και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 ερευνητικά πλοία τα οποία δεν έχουν καμία προστασία. Και χθε κάποιος μου είπε ότι προβλέπουν ε, όντως να προστατεύσουν και αυτά τα πλοία, δεδομένου ότι τα πλοία αυτά τα οποία είναι, έχουν ε, αναγνωριστική δραστηριότητα μπορούν ε, επίσης να τύχουν επιθέσεων. Αυτό αφορά τον αλληλευτικό στόλο, όπως σας είπα. Αυτό το οποίο είναι γεγονός είναι ότι η αύξηση των πειρατικών επιθέσεων προς το τέλος του έτους οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα τα πλοία τα οποία προστατεύονται πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν τα ψάρια. Στην ανοιχτή θάλασσα δηλαδή, εκεί που οι πειρατές κόβουν βόλτες. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση των αντιπυρατικών δυνάμεων. Από τις διάφορες ε, πληροφορίες τις οποίες έχουμε εμείς και βεβαίως πιο συγκεκριμένες πληροφορίες έχουν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης Αταλάντη, τι ξέρουμε όμως εμείς, ότι περίπου στον κόλπο του Άντεν υπάρχουν περίπου 20 στρατιωτικά πλοία και υπάρχουν και 6 περίπου στην Σομαλία, 4 βορείως των Σέιχελών. Ποια είναι η συμπλατική μου παρατήρηση, ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με κοινοτικά μέσα, στα πλαίσια της επιχείρησης Αταλάντης, αλλά λογικά πρέπει να πω ότι όταν ε, δραστηριοποιούνται, όταν γίνει προσπάθεια προσέγγισης από τους πειρατές ενός πλοίου της δικής τους ε, εθνικότητος. Μπορώ επίσης να πω ότι στην περίπτωση της Αλκανάρα ε, δραστηριοποιήθηκαν τα πλοία τα ισπανικά, για ένα γερμανικό τα γερμανικά, ένα εστιοφόρο αγγλικό ε, έγινε αντικείμενο πειρατεία και μία φρεγάτα αγγλική πήγε να βοηθήσει. Ποια είναι τα μέτρα τα στρατιωτικά που έχουμε. Αυτά που σας εξήγησα, αλλά πολλές φορές μειώνεται η αποτελεσματικότητα εξαιτία αυτού του παρατηρηθέντος μέχρι τώρα φαινομένου ο καθένας να βοηθάει τα πλοία της χώρας του. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και αεροπλάνα από τη Γαλλία, την Ισπανία, το Λουξεμβούργο και σύντομα μη επανδρομένα αεροσκάφη αμερικανικά. Και βεβαίως υπάρχουν διάφορες συνεργαζόμενες δυνάμεις στα πλαίσια της Αταλάντα, του ΝΑΤΟ, της Κίνας, της Ρωσίας, της Ιαπωνίας που μας βοηθούν. Έχουμε λοιπόν κάποιες ομάδες οι οποίες εξασφαλίζουν την προστασία. Φαίνεται ότι είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε για να προστατεύσουμε τα πλοία αυτά, τα οποία λιεύουν σε αυτές τις περιοχές, τα οποία είναι πολύ ευάλωτα, τα οποία δεν είναι πολύ ψηλά και τα οποία μένουν κινητοποιημένα για ώρες ή για μέρες. Αυτή είναι η λύση που εξευρέθη για να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα της επίθεσης. Απ' την άλλη πρέπει να πω ότι η επιχείρηση Αταλάντη, που πραγματικά είναι επιχείρηση προστασίας, είναι περισσότερο επιχείρηση συλλογής μυστικών πληροφοριών και αστυνομικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή με τον συντανισμό των δυνάμεων και με την ενημέρωση γίνονται ανιχνεύσεις βοήθεια από του, τα εναέρια μέσα για να γίνουν συλλήψεις πειρατών. Όλο και πιο σημαντικές και γρήγορες γίνονται οι συλλήψεις των πειρατών τελικά. Τα δύο συστήματα ή τουλάχιστον η... το ότι Γάλλοι συμπεριλαμβάνονται στην Αταλάντη οδήγησε σε καλύτερο συντονισμό όλων των προσπαθειών πρέπει στο μέλλον να δούμε πώς θα μπορέσουμε το σύστημα αυτό να το κάνουμε πιο ενοποιημένο και πώς θα μπορέσουν να συντονιστούν επίσης και οι δραστηριότητες των ε, ιδιωτικών ε, ιδιωτικού τομέα συστημάτων προστασίας. Τι θέλουμε κυρίως να αποφύγουμε οποιαδήποτε επαφή με τους πειρατές, να έχουμε πολύ καλή ενημέρωση για τις ενδεχόμενες δραστηριότητες τους και να μπορέσουμε σε περίπτωση προσπάθειας επίθεσης να αντιδράσουμε ταχύτατα. Εμείς ευθύς εξ αρχής υπογραμμίσαμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από την ροή πληροφοριών. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ καλή ροή μεταξύ των καραβιών της, ε, του ναυτικού, του γαλλικού και των υπολείπων μέσων που διαθέτουμε στην Επιτροπή. Τώρα, μίλησα για ενημέρωση. Είπα ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ε, προειδοποίησης. Υπάρχουν όμως προειδοποιήσεις οι οποίες γίνονται μετά από 4-10 ώρες και για ένα αλλιευτικό σκάφος είναι άχρηστο αυτό. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να μην τρενάρουμε. Πού οφείλεται αυτό το τρενάρισμα. Πρέπει να γίνει επαλήθευση στοιχείων από τον ε, στρατιωτικούς. Προτείναμε λοιπόν στα πλαίσια της Αταλάντης όποιες προδιοποιήσεις προέρχονται από τη λεκάνη Σομαλίας και κυρίως από τα αλλιευτικά σκάφη που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις ζώνες αυτές και ξέρουν πολύ καλά τι κάνει όποιο πλοίο περνάει από εκεί, πρέπει να διαβιβάζονται συστηματικά παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επαληθευθεί επισήμως. Πράγμα που θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία προειδοποίησης. Επίσης, το επίπεδο ταλάντης πρέπει να πω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ σαφές πρόγραμμα ταυτοποίησης των αλλιευτικών σκαφών. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιοι αλλιεύουν, είναι, ε, ποια ε, σκάφη είναι ευάλωτα, ποια είναι σε τράνζιτ, μόνο περνούν. Επίσης, ποια είναι τα πιο ευάλωτα πλοία. Τα πλοία του εμπορικού στόλου και τα αλλιευτικά. Και Όποιο και να είναι το μέγεθος, η ταχύτητα, η σημαία του πλοίου, θα πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί. Όταν λοιπόν γίνει η ταυτοποίηση πρώτα απ' όλα των αλευτικών στόλων, μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα πρέπει να κάνει για να διευκολύνει ε, την ροή πληροφοριών για να προστατεύσει αυτά τα πλοία. Σε επίπεδο Αταλάντης γίνεται ό,τι είναι δυνατόν ώστε οι νομικές πτυχές της μεταχείρισης των πειρατών να διευθετηθούν. Διότι έγιναν πολλές συλλήψεις πειρατών που κατέληξαν στην ε, ελευθέρωσή τους τελικά. Διότι όταν οι πειρατές βλέπουν να τους συλλάβουν, πετούν τα όπλα τους στη θάλασσα και το μόνο που μπορούν να κάνουν οι στρατιωτικοί είναι να τους στείλουν πίσω στη Σομαλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως εντοπίστηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε πειρατικές επιθέσεις και ακολουθήθηκε άλλη οντό. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω και που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τύχει προσοχής και από τα ενδιαφερόμενα κάτι αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα προσαρμόσιμο και μακροχρόνια σύστημα προστασίας. Ένα σύστημα λοιπόν ευέλικτο. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός των στρατιωτικών δυνάμεων και καλύτερη ένταξη όλων των συνιστοσών στην ε, πλαίσια του συστήματος επιχείρησης Αταλάντης. Είναι πολύ πολύπλοκες οι λύσεις. Δεν είμαστε κοντά τους. Κάποια από αυτά που επιθυμούμε παραμένουν προς το πάνω ευσεβείς πόθη, αλλά το να πιστεύει κανείς ότι με πολιτικά και διπλωματικά μέσα θα επιλύσει το πρόβλημα της πειρατείας επίσης είναι κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ εσάς. Κάποιος ευρωβουλευτής θέλει να παρέμβει. Ο κύριος Ρωμέβα παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη επιπλέον, διότι καθυστέρησα και δεν ήθελα να παρέμβω εγώ πρώτος, αν άλλο ήθελα να παρέμβουν. Όμως για μια ερώτηση ζήτησα και ίσως ε, ήθελα να την διατυπώσω. Ίσως ε, υπήρξε η τοποθέτηση, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω. Σε περίπτωση της προστασίας, ποιος είναι υπεύθυνο για αυτήν και με βάση την εντολή ποιο είναι υπεύθυνο για αυτήν την προστασία και υπό ποιου όρου και προποθέσει συγκεκριμένα σκάφη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αυτή την προστασία. Και εξηγώ τι γίνεται με ένα σκάφο που είναι ιδιοκτησία μια επιχείρηση που έχει την έδρα τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαία, α το πούμε, τρίτη χώρα ε, των Σιχελών του Παναμά, σημαία άλλη ε, οποιασδήποτε από το νομικό πλαίσιο, υπό το νομικό πρίσμα υπάρχει κάποια, ας το πω έτσι, περιορίζει το, τις δυνατότητες προστασίας που μπορούν να παρασχεθούν ή όχι. Δεν ξέρω αν είναι σαφές. Με ακούτε, με παρακολουθείτε. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, διότι πιστεύω ότι ε, υπήρξε κάποια, μια και υπήρξε διακοπή. Υπό το νομικό πρίσμα είναι το ερώτημα. Σε ένα σκάφος που είναι ιδιοκτησία μιας επιχείρησης που έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όμως έχει σημαία μιας τρίτης χώρας, ε, των Σεχελών του Παναμά, Ταϊβάν ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, υπάρχει περιορισμός ε, ο όρος περιοριστικός, η οποιασδηποτε άλλη χώρα. να δοθεί αυτού του είδους η ασφάλεια σε αυτό το σκάφος από πλευρά των Ευρωπαίων, των Ευρωπαϊκών Αρχών. Παρακαλώ. Λοιπόν, λέει η Πρώτα θα δώσω τον λόγο σε όλους και μετά θα πάτε εσείς τον λόγο να απαντήσετε. Εσείς παρακαλώ τώρα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να πω και να κάνω είναι να ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση, την εισαγωγή του εκπροσώπου του τομέα που θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένα θέμα πολύ μεγάλη ευαίσθησης, ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα αυτή τη στιγμή και επιπλέον ζούμε δραματικά την απαγωγή ενός ισπανικού πλοίου μέσα σε αυτό το πλαίσιο και υπάρχει μεγάλη ανησυχία των πολιτών για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Εγώ από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, δεν ξέρω αν κάνω λάθος ότι ότι είναι 45 περίπου σκάφη, έκανα πρόσθεση, 45 αλληλευτικά σκάφη που λειτουργούν σε αυτή τη ζώνη και αφορώνται 30 στρατιωτικά πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού και που εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις ε, και με την ε, συμμετοχή αεροπορικών μέσων ε, υπερπτήσεων κτλ. Είναι ένα θέμα αρκετά σύνθετου χαρακτήρα και πολύ περίπλοκο και σε σχέση με τις πληροφορίες, συλλογή πληροφοριών, τον συναγερμό, σίγουρα είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά για την, κατά, κατά των πειρατών πρέπει να είναι κανείς ταχύτατος και στη δράση του άμεσος και πρέπει να δοθεί άμεση απάντηση και με άμεση αντίδραση. Αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το ότι ταυτόχρονα τα προβλήματα που είναι τα αίτια της πειρατείας είναι αρκετά περίπλοκα και σύνθετα και αυτά απαιτούν μια απάντηση πιο ε, μακροπρόθεσμη και πιο σύνθετη γιατί ξεκινούν τα αίτια της πειρατείας ε, στην ε, ξηρά με τα προβλήματα της φτώχειας και της υπανάπτυξης. Πολύ περιπλοκά θέματα και επιπλέον τα προβλήματα που θέτουν απαιτούν μια διαφρομένη απάντηση, δομημένη όχι σε επίπεδο κρατικό μόνο, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε αρκετά συστηματικοί και συντονισμένοι. Και επιπλέον έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στη Σομαλία σήμερα, αλλά επίσης και σε διεθνές επίπεδο. Το πρόβλημα είναι μπορούν να υπάρχουν νόμιμες δραστηριότητες, ας σε διεθνή ύδατα τρίτων χωρών τέτοιου, είδους, τέτοιου χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο και σύνθετο. Θα ήθελα να ξέρω από πλευρά τη διάγνωση αυτή τη συνθετότητα και πολυπλοκότητα, αν υπάρχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένη εξειδικευμένη πρόταση, που ο τομέα θεωρεί ότι εμεί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, τα πρώτα μου λόγια θα είναι θα τα αφιερώσω στα άτομα εκείνα τα οποία έχουν απαχθεί στο πλοίο Αλακράνα, στο σκάφος αυτό, στους οικείους τους, στους συγγενείς τους και στους εφοπλιστές. Είναι κάτοικοι της δικής μου περιοχής και είναι γνωστοί και γνωρίζουμε και τις οικογένειές τους. Θέλω λοιπόν μετά από αυτό να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του γαλλικού τομέα της Γαλλίας για όλα όσα μας εξήγησε. Είναι γνωστή η αύξηση των επιθέσεων που υφίστανται κυρίως τους τελευταίους μήνες. Κάποιες επιθέσεις που είχαν προαναγγελθεί, προαναγγελόντουσαν από πλευράς του τομέα, που ζητούσε ο τομέας κατεπήγοντα μέτρα να ληφθούν για την προστασία του. Και είδαμε πως η Γαλλία έθεσε από την πρώτη κιόλα στιγμή τους στρατιώτες της, τους τοποθέτησε σε σκάφη με γαλλική σημαία. Δεν συνέβη το ίδιο με τα σκάφη με ισπανική σημαία, που ακόμα σήμερα βλέπουν και ζουν και βιώνουν πώς θα πρέπει με ιδιωτικούς ε, φρουρούς να προστατεύονται τα σκάφη της, ε, με ισπανική σημαία. Τούτο, λεχθέντο θα ήθελα να ξέρω αν με αυτή την εμπειρία που έχουν τα γαλλικά σκάφη με εκπροσώπους των στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας Πώς εσείς αξιολογείτε την ένταξη ιδιωτικών φρουρών στα σκάφη με ισπανική σημαία. Εσείς το αξιολογείτε με τον ίδιο τρόπο με, αυτό το οποίο πράττουν ως έργο επαγγελματίες στρατιωτικοί που από πλευράς ικανότητας και εκπαίδευσης και κατάρτισης η στρατιωτική αυτή είναι η μόνη εγγύηση για αυτά τα σκάφη, η μόνη εφικτή και αποτελεσματική εγγύηση. Κατά δεύτερο λόγο, θεωρείται επαρκές επιπλέον πέρα από τις προσπάθειες που μπόρεσαν να κάνουν οι χώρες στην ε, στο εγχείρημα Αταλάντη. Θεωρείται επαρκές ε, αυτό το οποίο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο γίνεται και έχει προβλεφθεί για αυτά τα σκάφη και με τα ελικόπτερα που δρούν εκεί και τα λοιπά. Και επιπλέον, τέλος, δεδομένων αυτών των τοποθετήσεων που ε, γινόντουσαν από κάποια μέσα του τύπου και από κάποιους εκπροσώπους, τουλάχιστον από πλευράς ε, της, Ισπανίας, της Ισπανίας, της ίδιας, πώς εσείς αξιολογείτε εκφράσεις ότι θα πρέπει να ψάξει να βρει άλλους αλευτικούς χώρους και τοποθεσίες ως, ε, μα. μας. Θα ήθελα να μου αξιολογήσετε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πραγματικά και είναι συνέπεια που απορρέει από συμφωνίες μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιπλέον ξέρουμε ότι αλλιεύουν και σε διεθνή υδατά. Αυτό απλά ώστε όλοι να μπορέσουν να γνωρίζουν το τι γίνεται με τις αλλιευτικές αυτές τοποθεσίες. Το θέμα δεν είναι απλό σε σχέση με τον ένα ή άλλο αλευτικό χώρο και περιφέρεια. Έχουμε λοιπόν αυτό το θέμα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπιλμπά. Η κυρία Νισμπαρέα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως βλέπετε είναι ένα θέμα που απασχολεί την Ισπανία σίγουρα όλους μας υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή τα δεινά τη επιπτώσει αυτή τη κατάσταση όλοι. Θέλω να διαφοροποιήσω κάπω το θέμα ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι ενό ε, σκάφου που αλλιεύει τόνου εκεί. Ε, δεν είναι θέμα καθόλου ισπανικό, είναι θέμα πανευρωπαϊκό. Είναι ένα θέμα που αφορά την ε, Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία αυτή τη στιγμή, γιατί τα σκάφη του αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη ζώνη. Και είναι ένα πρόβλημα γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα μορφή εγκληματικότητα, με αυτή τη μορφή πειρατεία αυτός πάρα πολύ πρέπει να ε, τύχει ε, της προσοχής μας και της αναγκαία, των αναγκαίων απαντήσεων. Αληθεύει και το είπε ο πρόσωπος του τομέα, ότι αυτό που κάνουμε είναι ψάχνουμε να βρούμε τα ε, ψάρια σε τα αλλιεύματα. Ξεπερνάμε δηλαδή γεωγραφικές περιοχές, ξεπερνάμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου υποτίθεται ότι υπάρχει εκεί εγγύηση για την ασφάλεια και απομακρυνόμαστε και προσπαθούμε εκεί να ψάξουμε να βρούμε τα αλλιεύματα. Πρέπει λοιπόν εδώ να λάβουμε υπόψη το θέμα και της ευθύνης. Όχι μόνο όμως το θέμα της ευθύνης. Αυτό δεν επαρκεί. Το θέμα της επίλυσης αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Το θέμα είναι διεθνούς χαρακτήρα. Έγινε λόγος για την αποτελεσματικότητα της δράσης Αταλάντη. Ήταν αποτελεσματική. Μειώθηκε σε αυτή τη ζώνη ο αριθμός των απαγωγών, παρότι αυξήθηκε σε άλλες περιοχές, σε άλλες ζώνες. Πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Ας πούμε ότι σε σχέση με στρατιωτικές δράσεις, σε σχέση με τους στρατιωτικούς ε, στα σκάφη, κάθε νομοθεσία κάθε χώρας επιτρέπει μια διαφορετική κατάσταση και δράση. Η Γαλλία έχει μια δυνατότητα με ενόπλους ε, ε, των ενόπλων δυνάμεων να διασφαλίζει τα σκάφη Η Ισπανία όχι. Είναι θέμα όμως και πρόβλεψης, προφύλαξης, πρόνοιας. Αναφέρθηκε ότι μια απάντηση στα αίτια πρέπει να δοθεί. Να βρούμε τα αίτια ποια είναι και να επανορθώσουμε να θεραπεύσουμε τις ρίζες του κακού και όχι το σύμπτωμα μόνο. Να ξεπεράσουμε δηλαδή τη στρατιωτική δράση απλά και μόνο. Σκέφτεστε να υπάρξουν διεθνείς σχέσεις, διεθνείς συμφωνίες αλληλεία που θα ρυθμίζουν και θα εξειδικεύουν με κάποιες συγκεκριμένες ρήτρε και ε, παραγράφους τι πρέπει να γίνεται σε σχέση με τέτοια θέματα και διπλωματικές δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων ώστε να μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα των σκαφών μια και είναι ένα πρόβλημα διεθνέ, το οποίο ξεπερνά το στενό πλαίσιο της Σα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Άνδρες Μπαρέ. Ο, η, κυρία Λεβίν παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτό το πρόβλημα άρχισε στη Σομαλία, όπως όλοι ξέρουν. Και πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα. Το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι από το 1991 δεν έχει κυβέρνηση η Σομαλία, δεν έχει ακτοφυλακή. Ε, δεν προστατεύει κανείς τα ύδατά της. Ε, διάβασα σήμερα μία συνέντευξη στο ίντερνετ με τον ε, υπηρεσιακό πρωθυπουργό, γιατί δεν υπάρχει ακόμη κυβέρνηση, και λέει αυτά που ακούμε συνήθως ε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ε, τα σχόλια που όλοι περιμένουν. Ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση και ότι έχουν ε, αλλιεύσει διάφοροι παράνομα στα ύδατα της Ομαλίας, Ευρωπαία Λύση και άλλοι. Και το έδωσαν ως δικαιολογία ότι έτσι άρχισε η Σομαλία άρχισαν να προστατεύουν τα ύδατά τους. Μαρκ λέγεται αυτός ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός και λέει ότι συνεχίζεται η παράνομη αλία στα ύδατα της Σομαλίας. και ε, αλλιεύονται ψάρια εκατοντάδων, αξίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ την ε, ημέρα. Ε, θα ήθελα να ακούσω κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μα αληθεύουν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ακούσουμε μία άποψη, μία τοποθέτηση για αυτό το σχόλιο. Μάλιστα. Βλέπω ότι ε, δεν ε, υπάρχει άλλο να ζητά τον λόγο. Θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Είναι σαφέ ότι αυτό που αποσαφίστηκε είναι το θέμα τη εναλλακτική λύση άλλων αλληλευτικών χώρων. Προφανώ κανένα από τα σκάφη που υπάρχουν εκεί, Ισπανικό, Γαλλικό ή άλλο. Δεν έχει κάποιο συμφέρον να ζει τέτοιες καταστάσεις και τέτοιο φόβο. Το λέω και το ξέρω αυτό. Υπάρχουν και μεγάλα σκαφή που όλοι βρίσκονται στους, ε, στις τραπεζαρίες και κοιμούνται εκεί διότι φοβούνται να μην υποστούν επίθεση. Λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν υπάρχουν άλλοι χώροι να αλλιεύει κανείς διότι τα διεθνή ύδατα έχουν ρυθμιστεί που μπορεί κανείς να ψαρεύει και που όχι. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί μια άλλη πορεία. Το θέμα είναι ότι η τροφοδοσία των ε, βιομηχανιών μας ε, με αλλιεύματα πάει εκεί ο, μας και πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος ε, το αλλιεύμα διότι σημαντικό ποσοστό της μεταπητικής μας βιομηχανίας το, το ψάρι, τα αλλιεύματα τα παίρνουν από τον Ινδικό και εδώ πρέπει να πούμε ότι 60% του ΑΕΠ των Σεϊχελών προέρχεται ακριβώς από τον πλούτο που παράγεται από τους δικούς μας ε, στόλους αληφτικούς εκεί και από τις δικές μας δράσεις. Υπό όλα τα πρίσματα λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχει ο στόχος της προστασίας αυτού του στόλου που βρίσκεται εκεί και που δεν έχει άλλες εναλλακτικέ λύσεις να ψαρέψει αλλού. Και οι άδειε είναι αυτές που υπάρχουν και οι δυνατότητες αυτές που υπάρχουν δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πολλοί πολιτικοί δεν θέλουν να το πούνε αυτό, αλλά είναι ένας τρόπος παραπλάνησης ε, των πολιτών. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά σε σχέση με τους ε, ψαράδες, τους αλείς. Το θέμα της Αταλάντης, της δράσης αυτής, είναι το θέμα της κοινοτικής δράσης που αποφασίστηκε στο άρθρο 1 για να έχει ως κύριο στόχο ανθρωπιστική βοήθεια και μετά προστασία των ευάλωτων σκαφών. Ευάλωτα σκάφη είναι τα εμπορικά πλοία και η αλληλεία πάντα θεωρεί, ε, θεωρεί το κάτι άλλο και κανείς δεν έδινε ιδιαίτερη προσοχή, διότι για αυτό το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν, η κοινοτική αλληλεία που υφίσταται εκεί, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια, ας το πω έτσι, ε, ιδέα ότι υπάρχει εκεί και δυνατότητα παράνομης ε, δράσης. Όμως ε, αυτό δεν, είναι, δεν αληθεύει. Να πει κανείς ότι σε σχέση με τέτοιες διεθνείς συμφωνίες μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επιπλέον ο Ινδικός ωκεανός ρυθμίζεται από μια περιφερειακή οργάνωση αλληλείας την OCTI και δεν είναι δυνατόν να πει κανείς ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους παρανομίες όπως κάποιοι ε, εικάζουν. Εδώ λοιπόν ε, σε σχέση με τη δράση Αταλάντη πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με τους υπεύθυνους που πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη εδώ θα ήθελα εγώ να πω το εξής. Εσείς είπατε πράγματι ότι η δράση Αταλάντη θα έπρεπε μέσω καλύτερων ελέγχων, καλύτερης δράσης και συντονισμού να προστατεύει τον αλληλευτικό στόλο εκεί και να προβλέψει με ειδικές δράσεις την κατάσταση αυτή. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη σε σχέση με τον κόλπο του Άντεν. Εμεί ε, συνεχίζουμε να εμένουμε και να επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει ε, επιπρόσθετη δράση. Όσον αφορά την ασφάλεια, υπάρχουν πεζοναύτες σε αυτά τα σκάφη. Πράγμα το οποίο τους βοήθησε πολύ να μπορούν έτσι με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν και να αποφύγουν επιθέσεις πειρατών. Όμως το θέμα είναι ότι άλλα σκάφη θα έχουν ιδιωτικούς φρουρούς, ιδιωτική ασφάλεια. Ιδιωτική ασφάλεια που σε ένα θέμα όπου το προσωπικό θα έπρεπε επαγγελματικά να έχει κατατιστεί και ε, προετοιμαστεί για τέτοιου είδους επιθέσεις. Και δεν είναι προετοιμασμένοι οι ιδιωτικοί φρουροί για τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Θα ήθελα να ξέρω σε σχέση με την ε, δράση Αταλάντη τι γίνεται. Θα προτιμούσαν οι στρατιωτικοί να έχουν απέναντί τους στρατιωτικούς, καταρτισμένου και εκπαιδευμένους και όχι κάποιους ιδιωτικούς φρουρούς με τους οποίους θα πρέπει να συνεννοούνται, που ιδιαίτερα στην ε, ισπανική περίπτωση πρέπει να είναι ισπανοί φρουροί και δεν έχουν ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ποια ασφάλεια θα δίνεται λοιπόν με τέτοιου είδου ιδιωτικού φρουρούς όταν έχουν απέναντί τους έναν πειρατή ή πειρατές. Ποιο είναι ο υπεύθυνο, ο εφοπλιστής του σκάφου, να συζητήσει με του στρατιωτικού για τέτοιε δράσει. Εφόσον υπάρχουν ιδιωτικοί φρουροί επί σκάφου, μπορεί να δημιουργηθούν πολύ σημαντικά προβλήματα και τριβέ. Δεν είναι ένα θέμα λοιπόν κόστου που πολύ εύκολα μπορούν να το αναλάβουν οι εφοπλιστέ και να το πληρώσουν, αλλά το θέμα τη ευθύνη. Ποιανού είναι η ευθύνη όταν έχουμε ευθύνη ενό ιδιωτικού φρουρού και υπάρξει κάποια, ε, ε, κάποιος φόνος ε, και σκοτωθούν άνθρωποι. Η δράση Αταλάντη, το εγχείρημα αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις πτυχές. Ξέρω ότι αυτές είναι αποφάσεις των κρατών μελών. Κάποια λαμβάνουν πιο εύκολα και καλύτερα τέτοιες αποφάσεις από ό,τι άλλα. Όμως πραγματικά υπάρχουν αυθεντικά προβλήματα με το να έχει κανείς ιδιωτικούς φρουρούς σε σχέση με τα σκάφη αυτά. Τούτου λεχθέντος θα πρέπει να εμείνω και να επιμείνω σε αυτό για το ότι η δράση Αταλάντη για άλλη μια φορά δεν έλαβε υπόψη συγκεκριμένες πτυχές ψυχέ για την, ε, τον αλευτικό στόλο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη και μάλιστα και σε σχέση με τον συναγερμό και την επιτήρηση. Θα ήθελα από πλευρά του εκπροσώπου να υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με την κοινή ακρόαση αυτό να ληφθεί υπόψη. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα ώστε να αντιμετωπιστούν εξάπαντο και να ξέρουμε αν μπορούν με αυτόν τον τρόπο να επιληθούν αποτελεσματικά. Καθώ κανεί δεν ζήτησε τον λόγο, εγώ παρενέβη ω τελευταία. Εσείς έχετε τώρα τον λόγο για να απαντήσετε σε κάποιες από τις ερωτήσεις που σα διατυπώθηκαν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήδη έχω απαντήσει σε διάφορα από αυτά τα ερωτήματα. Ας τα πάρω με τη σειρά. de savoir si on pouvait pêcher. Euh. Ε, το ερώτημα της κυρίας Μπιλμπάο. Αν μπορούμε να αλλιεύσουμε αλλού. Ναι, μπορούμε να στείλουμε αλλού τα σκάφη μας. Αλλά δεν έχουμε χώρο. Αφήστε που χρειάζεται και άδεια για να πάμε σε άλλα ύδατα. Στον Ατλαντικό έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Δεν μπορούμε να στείλουμε και σκάφη. Για τον Ειρηνικό πρέπει θέλουμε άλλη άδεια. Τέσσερις ευρωπαϊκές άδειε υπάρχουν για τον ειρηνικό. Τα σκάφη μας λοιπόν θα ε, ήταν υποχρεωμένα να λιεύουν ε, αν γινόντουσαν δεκτά στις διάφορες οικονομικές ζώνες μόνο σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή πρέπει να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους ε, δύο σκάφη. Παραδείγματο χάρη μπορούν να πηγαίνουν λέμε να στείλουμε δύο σκάφη μόνο, τα υπόλοιπα πρέπει να σταματήσουν. Για τις Αιγέλες, όπως σωστά είπε η βουλευτής, ε, πάει να πει ότι θα εκλείψει το ε, ίμιση του εισοδήματος, ακόμα και προσωρινά. η ασιατική βιομηχανία θα ε, κατακτήσει αυτό το μερίδιο της αγοράς αν επιστρεπτεί. Δηλαδή θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά αν φύγουμε από τον Ειρηνικό, ε, θα κροτηριάσουμε τον Ευρωπαϊκό Στόλο, ε, όχι κατά 40 σκάφη όπως ακούστηκε ίσως, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά πολλά σκάφη και θα εγκαταλείψουμε τους εταίρους μας από τη Μαδαγασκάρη, από τις Αιχέλες, από τον ε, Μαυρίκιο και θα τους αφήσουμε στην, ε, στο κακό πεπρωμένο τους. Μπορούμε να πάμε μόνο στον Ανατολικό Ειρηνικό. Μόνο εκεί. δεν σηκώνει πολλά αλλιεύματα, ε, έτσι είχε κατάσταση πάντοτε και αν δείτε και τους χάρτες ε, που ε, υπήρξαν οι επιθέσεις των πειρατών, ε, οι ζώνες ε, επικαλύπτονται με τις ε, αλλιευτικές ζώνες και αυτό ισχύει και στις Σεϊχέλες. Τι σημαίνει αυτό. Όπου και να πάνε στον ειρηνικό τα σκάφη για να γυρίσουν στις Σεϊχέλες διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιτεθούν οι πειρατές. Ούτως ή άλλως. Ακόμη και αν πάνε αλλού να αλλιεύσουν δεν γίνεται. Οι ναυτικοί μας οι... μας λένε όταν πάμε στο κανάλι της Μοζαμβίκης ή στη θάλασσα του Αργός. Χρειάζονται στρατιωτικοί γιατί θα μας επιτεθούν όταν γυρίζουμε. Αυτά για να δώσω μια πληρέστερη απάντηση. Ε, ε κυρία Λεβίν, Ε, ακούστηκαν αυτοί οι ισχυρισμοί για την ε, παράνομη αλληλεία. Για να σας απαντήσω θα έλεγα ότι μπορεί να είναι Σομαλή, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Ε, έπεσα πάνω στην ομιλία ενό ακαδημαϊκού από την Αφρική πρόσφατα που ανέφερε αυτό το επιχείρημα ότι σώζουν την αλληλεία οι Σομαλοί πειρατές. Για να σε εξηγήσω, για να καταλάβουμε καλά. Την περασμένη εβδομάδα έγινε ειδικό εργαστήρι για την μεταρρύθμιση το 2012 της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Ε, είχαμε ρετούς, ε, εκπροσώπους ε, των ΜΚΟ, εκπροσώπους των συνδικάτων, εμπειρογνώμονες, πλειοκτήτες. Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι η, τροπική, η αλία στους τροπικούς τηρεί τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, τις, ε, τα κοινωνικά πρότυπα, τα πρότυπα ασφαλείας, ε, σε βαθμό που στην πράσινη βίβλο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει την ερώτηση «Υπάρχει υποδειγματική αλία» δεν ξέρουμε, βρισκόμαστε σε αμηχανία, γιατί τελεαζόμαστε να πούμε «Ναι, η δικιά μας», αλλά δεν μπορούμε και να περηφανευόμαστε, έτσι. Ε, ξέρετε, υπάρχει ο συνασπισμός ε, για την ισότιμη αλληλεία και δεν σας μιλώ εδώ μόνο για την άναρχη αλληλεία, μιλώ για την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων κτλ. κτλ. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Δεν ισχύει, ε, δεν ισχύουν αφελίας. Και κάνουμε και συγκεκριμένε προτάσεις για να εκριζώσουμε αυτή την παράνομη αλία, γιατί και εμεί θύματα είμαστε στον Ελληνικό ωκεανό. Εκτιμούμε ότι 10% ε, των ε, αλλιευμάτων κάποιων ειδών αντιστοιχούν στην παράνομη αλία ε, και ζητούμε την απαγόρευση της μεταφόρτωσης εμπλό. εξαρτάται βέβαια γιατί δεν γίνεται σε κάποιους, με κάποιους τόλους ούτως ή άλλως. Έχουμε το VMS, έχουμε το ηλεκτρονικό ημερολόγιο, το ημερολόγιο μάλλον, ε, ορισμένες φορές ε, ε, έχουμε και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πάνω στα σκάφη. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστούμε αυτό που κάνουμε. Και για να απαντήσω και στον κύριο Σάντσες, θα έλεγα ότι θα θέλαμε να ζητήσουμε το εξής από το Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με, να ε, με μεγαλύτερη πυγμή, με πιο αυστηρό τρόπο να ε, ε, επιμείνει ότι είναι νόμιμη η αλληλεία της σε ύδατα τρίτων χωρών και συγκεκριμένα στον Ειρηνικό ωκεανό στη λεκάνη της Σομαλίας. Γιατί δεν έχουμε τόσο άλλο αλληλευτική συμφωνία με Σομαλία. Δεν μιλάω για τα σομαλικά τι μιλάω για τα διεθνή στην λεκάνη τη Ο κύριος Δρομέβα τώρα, ε, τι, τι ακριβώς με ρωτήσατε. θα απαντήσει μάλλον ο συνάδελφός μου στην ερώτηση του κυρίου Ρομέβα. Ναι, μιλήσατε για ιδιωτικές φρουρές. Εξαρτάται από τη σημαία, από το κράτος σημαία και από τη δική του νομοθεσία. Ε, να κάνω μια αντιπαραβολή ανάμεσα στην Ισπανία και στη Γαλλία για να καταδείξω ότι κάποιες νομοθεσίες προβλέπουν παρέμβαση στρατιωτικών, άλλες όχι πάλι. Θα προσθέσω και κάτι άλλο γιατί ακούστηκε στι ερωτήσεις ότι από την εμπειρία μας ε, προτιμάμε εμπλό να υπάρχουν στρατιωτικοί και όχι ιδιωτικέ φρουρές γιατί έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και έχουν συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις παρεμβάσεις τους. Ε, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος ε, και ελπίζω να μην ε, υλοποιηθεί αυτό. Να υπάρξουν κάποιοι που εγώ τους ονομάζω cowboys. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα σκάφη μας και τα πληρώματά τους, αλλά δεν πάμε να κυνηγάμε τους πειρατές, ε. Αν μια ζώνη θεωρείται άκρος ε, επικίνδυνη βάσει των πληροφοριών παίρνουμε από ε, το ναυτικό, ε, η πρώτη εντολή είναι να φύγει το σκάφος από τη ζώνη για να μην υποβληθεί σε αυτό το κίνδυνο. Δηλαδή η πρώτη άμυνα είναι η φυγή. Μόνο όταν σε κατάσταση άμυνας οι στρατιωτικοί που είναι θα παρέμβουν βάσει αυτού του πολύ συγκεκριμένου ε, πρωτόκολλου για να μην κλιμακωθεί η ένταση. Μόνο σε κατάσταση ε, άμυνας. Και φυσικά, πάση θυσία, αποφεύγουμε να ε, ανέβει ο πειρατής στο σκάφος, γιατί αλλιώς έχουμε χάσει το παιχνίδι. τώρα, αυτό δεν προβλέπεται στην Ισπανική νομοθεσία, είτε μιλάμε για την προστασία του σκάφους, είτε του πληρώματος. Και γι' αυτό προτείνεται η χρήση αυτών των ιδιωτικών ε, φρουρών. Ευχαριστούμε κύριε Βέρ. Νομίζω ότι με αυτή τη τελευταία απάντηση εξαντλήσαμε τα ερωτήματα. Υπάρχει ένα γενικό ερώτημα που θέσατε και εσείς Πρόεδρε. Δηλαδή, αν η επιχείρηση Αταλάντη Ε, συνιστά επαρκή απάντηση στα, για τα προβλήματά μας. Η Αταλάντη, η διάσταση της επιχείρησης δεν ε, μπορεί να καλύψει τα λιευτικά σκάφη. Ε, αν ε, ούτε και φτάνει ε, να έχουμε τους στρατιωτικούς εμπλό. Χρειαζόμαστε ανάντι και αστυνομικούς στην ξηρά. Ε, τα μέσα της επιχείρησης πολλαπλασιάζονταν. Έχουμε δύο φρεγάτες που αυτό αντιστοιχεί σε 300 άτομα, αν δεν κάνω λάθος με μία φρεγάτα και με ένα και μία ομάδα στρατιωτικών σε κάθε σκάφος του στολίσκου με 150 στρατιωτικούς ε, δηλαδή με λιγότερα άτομα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι αν είχαμε δύο φρεγάτες. Η προστασία εν πλώ μας επιτρέπει οι στρατιωτικοί άμεσα να ξέρουν ε, τα πάντα για τις επιθέσεις των ε, πειρατών ε, και μπορούν να γίνουν και ταχύες επιχειρήσεις των αστυνομικών της ακτοφυλακής. Είναι συμπληρωματική η δράση. Πάλι ευχαριστώ. Πολύ σύντομα πάλι ζήτησε λόγο ο κύριος Ρόμεβα. Σε σχέση με το θέμα της σημαία, εάν κατάλαβα καλά, από την απάντησή σας. Η σημαία του πλοίου καθορίζει την δυνατότητα να έχουμε στο σκάφος στρατιωτικούς. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, παρά το γεγονό ότι πρόκειται για επιχειρήσει ευρωπαϊκές, εάν δεν έχει ένα πλοίο ευρωπαϊκή σημαία, δεν μπορεί να τύχει προστασία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όσον αφορά τους στρατιωτικούς που βρίσκονται Καταλάβατε απολύτως τι είπα προηγουμένως. Εξαρτάται από την κατάσταση της σημαίας του πλοίου, του κράτους, δηλαδή της σημαίας του πλοίου οι παρεμβάσεις των στρατιωτικών δυνάμεων στον κόλπο του Άδεν και στην Σομαλία πρέπει να πω ότι γίνονται στο πνεύμα της αλληλεγγύης. Εάν ένα αλληλευτικό σκάφος, το οποίο δεν είναι αλληλευτικό σκάφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δυσκολίες και είναι πολύ κοντά του ένα πολεμικό πλοίο, χωρίς να μπορώ να το ορκιστώ, σίγουρα σχεδόν θα μπορούσα να πω ότι θα πάει να βοηθήσει. Η Αταλάντη παρά την πραγματογνωμοσύνη της και τα μέσα που διαθέτει, δεν είναι εξειδικευμένη στην προστασία ληφτικών στόλων. Η Αταλάντα, η Αταλάντη, συγγνώμη, αν θέλετε, παίζει το ρόλο της αστυνομίας στην περιοχή. Και επειδή ξέρουμε πώς επιτίθενται, δεν έρχονται ούτε με βαρκάκι ούτε με κανό. Ανατρία τα σκύφ φτάνουν. Και τα μικρά, τα σκύφ δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει το ραντάρ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε πολύ γρήγορο χρόνο μπορούν να επιτεθούν σε ένα πλοίο. Εάν τώρα έχουμε μεγαλύτερα σκάφη, μπορεί κανείς να κάνει καλύτερα τη δουλειά του για να εξακριβώσει εάν πρόκειται για πλοίο πειρατικό ή κάποιο άλλο αλληλευτικό σκάφος. Δεν μπορώ να πω ότι όποιο περνάει και δεν είναι δικός μας από εκεί είναι πειρατής. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει η Αταλάντη και με ένα αέρια μέσα και με την είδους αυτή την αστυνομία του ρόλο τις οποίες παίζει η Αταλάντη και με άλλα σκάφη τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον ελευτικό μας τόλο. ευχαριστώ. Μια σύντομη ερώτηση θα είχα πόστα. Τι γίνεται αν ας πούμε συλληφθούν πειρατές Ποιες ποινές ε, θα επιβληθούν από πλευράς ε, ε, κρατών. Είναι αυτό αποτρεπτικό ως ποινή ή οι μικρέ ποινέ ε, είναι, α το πω έτσι, κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Μπαρέα. Θα ήθελα μία διευκρίνηση για την ερώτηση που έκανα προηγουμένως για τις, τα προληπτικά μέτρα. Προβλέπετε κάποια ε, μέτρα ειδικέ συμφωνίες, ειδικέ ρήτρε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα πειρατείας για να όλα προβλέπονται από την περιοχή εκείνη. Μας λέτε ότι όντως η επιχείρηση Αταλάντη έχει καταλήξει θετικά αποτελέσματα, δουλεύει το σύστημα και θα πρέπει να την ενισχύσετε. Ε, πιστεύετε ότι εάν ε, κάθε κράτος εφαρμόζει ρητά την ε, δική του νομοθεσία, οι δικασίες που προβλέπονται θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της Αταλάντης. Θα ήθελα να πω σε ε, οποιοδήποτε από εσά ότι εγώ δεν απάντησα προηγουμένως, όπως είπατε σε κάποιες ερωτηστικές σα απλώς έκανα και εγώ κάποιε παρατηρήσει. Έχετε το λόγο. Ορίστε, κυρία Βουλευτά, ξέχασα κάπω την ερώτηση που υποβάλλατε. Και έτσι θα απαντήσω και στην κυρία Ρόρνταστ. Εγώ δεν είμαι νομικός, θα σας δώσω κάποια στοιχεία, αλλά κυρίως αφορά ένα νομικό η ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι σήμερα οι περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν την κατάλληλη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουν από νομική σκοπιάς τις ε, πειρατικές επιθέσεις. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή οι γερουσιαστές μας και οι βουλευτές μας εξετάζουν νομοσχέδιο για την ε, διευκόλυνση της δράσης των ε, στρατιωτικών μας για να μπορέσουμε να εκριζώσουμε τα φαινόμενα πειρατείας. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν ε, οι συμφωνίες της Montego Bay που θα πρέπει να αποτελέσουν το υπόδειγμα και να δούμε πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στα πλαίσια κάθε εθνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν οι ακτοφύλακες από τις Σεϊχέλες σχεδόν συνέλαβαν πλοίο πειρατών που είχαν επιτεθεί στους Γάλλους, ο δικαστής από τις Σεϊχέλες, σύμφωνα με το δικό του σύστημα, αποφάσισε να τους ε, στείλει στη χώρα τους ελεύθερους, να τους ελευθερώσει τους στη χώρα τους διαφορετικά αν τους είχε φυλακίσει, είχε κάτι κάτι άλλο, κάποιος ε, ε, δικηγόρος θα μπορούσε να τους υπερασπιστεί ισχυριζόμενος ότι υπάρχει νομικό κόλλημα. Βάσει λοιπόν των συμφωνιών του Μοντέγο Μπέι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό, ότι δεν είμαι νομικός. Πρόκειται λοιπόν για μία της που να καταβάλουμε σήμερα, αλλά δεν μπορώ να σας πω εάν πρόκειται για κάτι το οποίο εξαρτάται από την Αταλάντη. Ίσως κάτι κοινοτικό, σε κοινοτικό επίπεδο, κάτι που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα εσάς, για να δείτε πώς με αυτές τις χώρες εταίρους στον Ινδικό ωκεανό θα πρέπει να κάνετε κάποιες διαβουλεύσεις σε διμερές πολυμερές επίπεδο ώστε να μπορέσει και η σχετική νομοθεσία του καθενός να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Για να τελειώσουμε, διότι τελειώνουμε, εγώ είμαι ευέλικτη, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα έχουν και κάποιο όριο. Κυρία Μπιλμπάο, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τη γενναιοδορία σας. Απλώς και μόνο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του κλάδο που ήθελαν, μας έδωσαν τις εξής και να πω, κάνω δύο παρατηρήσεις. Στην τελευταία σαν της Επιτροπής είχαν πει κάποιοι αλλοίς ότι η επιχείρηση Αταλάντη δεν είχε ως στόχο την προστασία των ευτικών σκαφών. Και με ένα ψηφισμό ζητήσαμε να επεκταθεί η προστασία εκτός των εμπορικών πλοίων και στα αλλιευτικά σκάφη. Εγώ πήρα μια απάντηση σε μια ερώτηση την οποία είχα υποβάλει το Σεπτέμβριο από το Συμβούλιο, δεδομένου μας ανησυχούσαν τέτοιου γεγονότα και θα διαβάσω μόνο μία παράγραφο, δεδομένου ότι πρόκειται για το θέμα που συζητούμε. Λέγει το Συμβούλιο λοιπόν ότι η απόφαση να προστατευτούν τα αλλιευτικά σκάφη που βρίσκονται ε, κοντά εκεί που ενεργούν εξαρτάται από κάθε κράτος μέλος. Άρα και η Αταλάντη και τα κρατημέλη έχουν ευθύνη και όπως λέει το Συμβούλιο εμπίπτει κυρίως η ευθύνη σε κάθε κράτος μέλος. Θα ήθελα εδώ να σας πω ποια είναι η θέση μου καθώς και η θέση του κόμματος και της ομάδας που εκπροσωπώ. Το κόμμα μου είναι το Εθνικό Νικιστικό Βασκικό Κόμμα. Ξέρουμε ότι αυτό το οποίο χρειάζονται τα λιευτικά σκάφη με ισπανική σημαία είναι να υπάρξουν στρατιωτικοί και επ' αυτών δεδομένου ότι είναι κάτι το οποίο έγινε για τους Γάλλους και ξέρουμε τώρα πρόσφατα ότι κάποια λιευτικά σκάφη δέχτηκαν επιθέσεις διότι όπως λέτε είναι πάρα πολύ πιο φθηνό το μέσο αυτό. Αν έχουμε σε μια φρεγάτα ε, του πολεμικού ναυτικού 300 άτομα που δεν μπορούν να προστατεύσουν, τι κάνουμε. Καλύτερα να έχουμε μικρές ομάδες σε κάθε σκάφος. σκάφος. Επαναλαμβάνω, είναι πιο αποτελεσματική αυτού του είδους η προστασία, πιο φτηνή και θα θέλαμε το μέτρο αυτό να επεκταθεί και στα ισπανικά αλληλευτικά σκάφη. Δεν δίνω σε κανέναν άλλο το λόγο. η κυρία Μπιλμπάου θα κάνει μια ερώτηση και κάνει ολόκληρη παρέμβαση. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι η Επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχει να πει. Ακούστε κύριε Σάντσε. Δύο φορέ πήρατε το λόγο. Είπα ότι τελευταίο συνάδελφο τον οποίο έδωσε το λόγο είναι η κυρία Μπιλμπάου. Πρέπει και εγώ να ενεργήσω πρόεδρο. Διαφορετικά τι κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του εκπροσώπου του τομέα Λυπούμε που δεν ήρθαν οι συναδελφοί. Εσεί κάνατε ό,τι μπορείτε για να μπορέσετε να εκπροσωπήσετε όλο τον τομέα, αλλά όντω ο καθένα έχει τα δικά του προβλήματα. Ο κύριο Καντέκ θα μα εκπροσωπήσει ω συμπρόεδρο αυτή τη κοινή ακρόαση που έχουμε με άλλε επιτροπέ. Θα επαναλάβουμε τα αιτήματα που έχουμε, δηλαδή η επιχείρηση Αταλάντη να τύχει ειδική μεταχείρισης όπως είπατε και εσείς, για να μπορέσει να γίνει κάτι για τον αλληλευτικό στόλο. Σας ευχαριστώ, καλή τύχη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι προσπάθειες μπορούμε ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρα στην αποστολή του η επιχείρηση Αταλάντη και αν μπορεί να επεκταθεί και στα αλληλευτικά σκάφη, διότι όπως είπατε και εσείς είναι σημαντικό και θα προσπαθούμε εμείς από τη θέση μας να παράσουμε την καλύτερη δυνατή βοήθεια. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων Ρέγκας στο δυτικό τμήμα τη Βαλτική θάλασσα. Η κυρία ρόντου και ο κύριο Σπούγκ ζήτησαν να παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας εξηγήσει την ειδική κατάσταση της Ρέγκας στο δυτικό τμήμα της Βαλτικής θάλασσας. Δίνω λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στην ε, Κομισιό ή σε εσάς. Ας λάβει το λόγο πρώτα λοιπόν η Κομισιό. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής λοιπόν. Μια στιγμή να δω ποιος είναι. Εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Συγγνώμη που δεν ε, γνωρίζω το όνομα. Έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ευχαριστώ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει την κατάσταση στην Βαλτική θάλασσα όσον αφορά την Ρέγκα στο δυτικό τμήμα της Βαλτικής. Η κατάσταση των αποθεμάτων εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρή. Υπάρχει μείωση σημαντική κατά από 15% σε 30% ετήσια από το 2004 και το 2008 αναμένεται να είναι το χαμηλότερο αυτό το απόθεμα και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα αναστραφεί αυτή η τάση στο εγγύς μέλλον. Λόγοι για αυτή την κατάσταση δεν είναι γνωστοί, για αυτή την φθήση παρέμεινε στο χαμηλότατο ιστορικό ποσοστό αυτό το απόθεμα τα τελευταία χρόνια και αναμένεται ακόμα περισσότερο ταχύτερα να συνεχίσει την φθήνουσα πορεία στο άμεσο μέλλον <clears throat> λόγω της ε, κατάστασης αυτής. Ταυτόχρονα η θνησιμότητα των ε, ηχθείων είναι πολύ υψηλότερη και το απόθεμα υπεραλλιεύεται. <clears throat> Υπάρχει σύσταση για την ε, μείωση ακριβώς της θνησιμότητας των ηχθείων το 2009 για να υπάρξει μια δραστική μείωση βιομάζας. Η μείωση αυτή κατά 31% για την βελτίωση των πραγμάτων. Όμως η Επιτροπή πρότεινε η ποσόστοση για τη ρέγγα στη Δυτική Βαλτική κατά 21% μόνο να μειωθεί η αλληλευτική προσπάθεια, λαμβάνοντας μόνο υπόψη τις οικονομικές ανάγκες των ε, επιχειρήσεων αλληλείας. Εμείς θεωρούμε ότι μια μείωση κατά 21% είναι ε, το ελάχιστο μέσο και μέτρο ώστε η θνησιμότητα των νυχθείων να μην αυξηθεί τουλάχιστον. Το απόθεμα ρεγγών που αλλιεύεται στην Δυτική Βαλτική και στην, στο Σκαβιεράκι και στην Κατεγάτη. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο διτό χαρακτήρα, το 22-24 και το 3α ως υποδιαρέσεις επιστημονική ε, συμβουλή σε σχέση με τα αποθέματα αυτά που υποκατανέμονται με βάση πολιτική συμφωνία στη συνάντηση του Συμβουλίου στο Λουξεμβούργο στις 19 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι η αλλιευτική πίεση επ' αυτών των αποθεμάτων δεν θα πρέπει να αυξηθεί. Μια αντίστοιχη μείωση των ΤΑΚ για το 2010 θα πρέπει εξάπαντος να είναι ισορροπημένοι με διαφορετικό τρόπο, διαφοροποιημένα. Τα τάκ για την Δυτική Βαλτική κατά 16,5% θα μειωθούν. Μόνο ενώ για τον Κατεγάτη και την Σκαγεράκη η μείωση θα πρέπει να είναι 25% που στοχεύουμε ως επίπεδο μείωσης. Τελικά ΤΑΚ για τις ε, περιοχές αυτές θα εξαρτηθούν φυσικά από τις διαπραγματεύσεις ως ήθιστε με την Νορβηγία και θα ληφθεί απόφαση το Δεκέμβριο και όχι νωρίτερα. Αυτό θα βοηθήσει να απαμβληθούν οι άμεσες επιπτώσεις στις ε, επιχειρήσεις και βιομηχανίες χωρίς καθυστέρηση χρειάζεται λήψη μέτρων που θα ρυθμίζει αυτές οι υποθέσεις ώστε να επιτραπεί στη βιομηχανία να προετοιμαστεί για τη μεσοπρόθεσμη μείωση των αποθεμάτων όπως αναμένεται. Γι' αυτό το στόχο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνατότητα πολυμορφοποίησης δραστηριοτήτων για την αλίευση, καθώς επίσης και μέτρα για την αναβάθμιση των αλλιευωμένων και εκφορτωνόμενων ποσοτήτων, καθώς μέτρα και μακροπρόθεσμα για την αλλιευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, Σα ευχαριστώ εσά Και στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο ο κύριος Κούν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής ακούσει ότι αυτό το είδος ρέγγας είναι διασυνοριακό και ότι η έδρα του είναι στη Σκαγεράκη και στο Κατεγάτη, δηλαδή στην είσοδο της Βαλτικής. Το νηπιαγωγείο βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της ε, Βαλτικής, στα ε, ριχά ε, νερά κοντά στη δική μου περιφέρεια. Και κατά τα τελευταία δέκα χρόνια και πιο πριν είχαμε και το θέμα το οποίο απαντήθηκε πιο πριν, πώς έχει η υγεία των αποθεμάτων αυτών και οι προτάσεις ίσες που έχουν υποβληθεί σε σχέση με την Επιτροπή και οι συστάσεις από αυτό το όργανο προς την Επιτροπή. Τώρα δεν είναι νέα λοιπόν μέτρα αυτά τα οποία εισάγονται ή υιοθετούνται, αλλά για την προστασία των αποθεμάτων. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε δραματικές μεταβολές και αλλοιώσεις των αλλιευμάτων που εισήχθησαν ως ρύθμιση και που μία εκ των βάθρων αλλαγή των στόλων που αλλιεύουν ρέγγα και στη Γερμανία και στην Δανία και στην ε, περιοχή αυτή της Βαλτικής. Αυτή ήταν η επίπτωση. Αν επιτρέπετε να παρουσιάσω τα αριθμητικά αυτά μεγέθη, το 1998 είχαμε τάκ ποσόστοση συνολικά 150.000 τόνων που μέχρι το έτος 2008 σε 21.000 τόνους ε, μειώθηκαν. Από 150.000 σε 21.000 τόνους. Τεράστια δηλαδή επέμβαση αυτή για όλους τους εμπλεκόμενους για να προστατευτεί το απόθεμα ρεγγών. Αυτό τι σημαίνει φυσικά. Σημαίνει μια δραστική μείωση του στόλου, του ε, αλευτικού στόλου. Το ακούσαμε και πιο πριν. Τα μέτρα που πέρσι μέσω της ΙΤΣΕΣ ε, για το 2009 συστάθηκαν ήταν 69% αυτών των 21.000 τόνων. Καθένας μπορεί να φανταστεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που δημιουργείται για τους αλληλείς μας, παράκτιους και μη, λόγω αυτής της κατάστασης. Και η οικονομική τους επιβιωσιμότητα βρίσκεται πραγματικά εν κινδύνο, διακυβεύεται πολύ σοβαρά. Και γι' αυτό κατά τούτο μπορώ να πω ότι είναι αναγκαίο λοιπόν εμείς σίγουρα με τις επιστημονικές αυτές, με τα επιστημονικά πορίσματα, αλλά από κοινού και με, τα, ράτς, με, τα, με τους κλαδικούς εκπροσώπους των αλλιέων να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Φυσικά είναι θλιβερό ότι κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει ακριβώς και ούτε οι δικοί μας επιστήμονες, ούτε οι αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Αυτό δηλαδή το απόθεμα ρεγκόν να έχει υποστεί μια τόσο σημαντική μείωση και να έχει συρρυκνωθεί τόσο πολύ Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γι' αυτό, πώς δηλαδή ε, εξελίχθηκε η βιομάζα των αποθεμάτων αυτών. Αυτή τη στιγμή η γόνη σε κάποιους τομείς είναι κατά 30% λιγότερη. Αυτό έχει αποδειχθεί. Αλλά στο τέλος τέλος δεν μπορεί να είναι μόνο αποτέλεσμα υπεραλίευσης αυτό. Αν δει κανείς ε, πώς έχει διαμορφωθεί η αλία και πώς αντέδρασε η αλία και από 150.000 τόνους πήγε σε 21.000 τόνους και μειώθηκε σημαντικά, ε, τότε αυτό πιθανώς έχει και βιολογικά αίτια ως κατάσταση. Γιατί εδώ έχουμε μια τόσο σοβαρή κατάσταση εις βάρος των ρεγκών. Και αυτά που από επιστήμονες αλλά και από αλληλείς ακούω και πληροφορούμε, πρόκειται για την βάση τροφής την ίδια την τροφή που χρησιμοποιούν οι Ρέγγες. Προτού αρχίσουμε να υιοθετούμε δραστικά μέτρα, ριζικά, ριζοσπαστικά μέτρα, πρέπει να βρούμε σε ποια, σε ποια αίτια οφείλεται για το ότι κατέληξε σε μια τέτοια κατάσταση το απόθεμα ρεγγών. Στην τελευταία περίοδο, αυτό μου είπαν οι παράκτη αλληλείς ρέγγας από την περιοχή μου, μου είπαν ότι εξαιρετικά λειτουργήσε η προσπάθεια. Επειδή όχι μόνο είδαν τα αποθέματα, αλλά και μπόρεσαν και να αλλιευθούν με τρόπο που δεν τα είχαν δει επί δεκαετίες. Ακριβώς όσον αφορά και το απόθεμα των ηλικιωμένων ε, ενήλικων ε, ηχθείων. Και με τις περιορισμένες ποσοστώσεις που τους είχαν εγκριθεί, σε λίγες μέρες είχαν αλλιεύσει το ποσοστό το οποίο τους είχε δοθεί και είχαν επιστρέψει. Και αυτά τα οποία περιφέρθηκαν και στην Γκράμπο και στην άλλη μου περιφέρεια ήταν τόσο καλά κατοικημένα από ε, ενήλικα ψάρια που υπήρχε δυνατότητα αλίευσης έντονα και πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε από επιστημονικά συμπεράσματα και πορίσματα αλλά και από την ίδια την πείρα και εμπειρία των αλλιέων να επικαιροποιήσουμε τις γνώσεις μας, να δούμε τι γίνεται και σε τι οφείλεται. Είμαι στη διάθεσή σας καθώς επίσης και οι συνάδελφοι από το Schleswig Holstein ώστε όλη την πείρα μας να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε, να αντλήσουμε συμπεράσματα για την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ εσείς κυρία έχετε τον λόγο κυρία Ρόντες. Είναι πολύ αξιόλογη η πρόταση του κυρίου Κούν, αλλά δεν είμαι εγώ η ικανή από πλευρά πραγματογνωμοσύνη για να κρίνω. Και στρέφομαι και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούμε ότι υπάρχει υπεραλίευση που έγινε τα τελευταία χρόνια. Σημαντική υπεραλίευση. Πρέπει να το δεχθούμε, θα έλεγα αυτό. Ακόμα και για την περίπτωση αν στην περιοχή Ρούγκεν είναι διαφορετική κατάσταση όπου είναι πολύ υγιής ας πούμε ο πληθυσμό ε, των αποθεμάτων. Αλλά πρέπει να δούμε σε σχέση με τη συνολική Βαλτική θάλασσα τι έγινε στις τελευταίες δεκαετίες. Υπήρξε πραγματικά έντονη υπεραλίευση. Όμως εδώ υπήρξε και προβλεπόμενη ανάκαμψη. Και τουλάχιστον αυτό μου είπαν επαΐοντες. Διαπιστώθηκε ότι τα ε, ψάρια τα οποία γέννησαν είναι διαθέσιμα, αλλά δεν υπάρχουν οι γόνοι, δεν υπάρχει επόμενη γενεά. Το ότι γέννησαν τα αυγά τους αυτά τα ψάρια, εντάξει, αλλά στη συνέχεια κάτι συνέβη και κανείς δεν μπορεί να το επεξηγήσει τι συνέβη, γιατί αυτά τα αυγά δεν οδήγησαν σε νέο πληθυσμό ψαριών. Μπορεί να οφείλεται σε οικολογικά προβλήματα, ρήπανση ή άλλα. Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες και οικοτολογία. Δεν υπάρχει καμιά ακριβής επιστημονική εξήγηση και ακόμα και αν σε σχέση με τη Βαλτική, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι η τροφή των ρεγγών δεν είναι η ίδια όπως ε, πριν από 50 χρόνια, δεν είναι της ίδιας ποιότητας και ότι στο πλανκτόν, ως δομή του πλανκτόν έχουν αλλάξει πάμπολα πράγματα. Αυτή δεν είναι η μόνη και αποκλειστική λύση. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς να δώσουμε την εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μια μελέτη που αυτό το φαινόμενο θα το εξετάσει σε βάθος, διότι πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα και για άλλα αποθέματα άλλων ψαριών η ίδια κατάσταση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ξαφνικά. Να καταλήξουμε ξαφνικά σε μια κατάσταση όπου τα αυγά δεν θα εποαστούν και δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει νέος πληθυσμός ψαριών. Είναι σαν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Κάτι πρέπει να υπάρχει πίσω από αυτή την κατάσταση και πρέπει να το ανακαλύψουμε, να το βρούμε. Ε, λοιπόν, αυτή την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε και να βασιστούμε σε αξιόπιστη στα στοιχεία, επιστημονικά στοιχεία για να βοηθήσουμε τους αλληλεί εν τέλει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρόντε. Ο κύριος Γκρόμπατσικ παρακαλώ. E, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε ε, η παράκτη να επαναπροσανατολίσουν ε, τις ε, δραστηριότητες τους για να αλλιεύουν ε, ρέγκα. Δύο χρόνια μετά, έκδηλα, πρόκειται για λάθος. Διαπιστώνουμε. Ευτυχώς δεν είχαν αλλάξει όμως τι δραστηριότητε τους, ε, γιατί πώς να χρησιμοποιήσουν τα δεκάμητρα σκάφη για να ψαρεύουν ρέγγα. Αν είχαν ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε αφοπλιστεί το σκάφος τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προτάθηκε επίσης να προστατεύσουμε το γάδο. Η, γιατί η Ρέγκα και η Σαρδελόρεγκα έτρωγαν τα αυγά του γάδου. Ήταν δηλαδή επιβλαβής οργανισμοί, μας έλεγε η Επιτροπή. Εδώ μιλάμε για την βιομηχανική αλληλεία και αναρωτιόμαστε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε ένα δίχτυ 18 μέτρων για να έχουμε ένα τεράστιο δίχτυ που καλύπτει όλη τη Βαλτική. Αλλιεύονται αυτά τα ε, ψαριά για να φτιαχτούν ηχθιάλευρα για να δοθούν στις ιδεατοκαλλιέργειες. δεν υπάρχει στρατηγική. Μιλήσαμε για την περιφερειοποίηση, για την προστασία ε, των ε, μικρών ε, ε, σκαφών. Τι θα κάνουμε λοιπόν, ε, θα ακολουθήσουμε την λύση που προτάθηκε για τις φώκες. Ας αρχίσουμε να πυροβολάμε τους κορμοράνους, δεν βλέπω άλλη λύση. Ίσως να πρέπει να πυροβολήσουμε και στους ίδιους τους ψαράδες. Ίσως αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Ε, πάντως αυτά είναι τα προβλήματα στη Βαλτική. Και άρα τι πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι η λύση. Μα είναι απλό. Χρειαζόμαστε ε, έρευνα με λογικά πορίσματα αλλά δεν επαρκεί αυτό. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλα τα είδη, το γάδο, τη σαρδελόρεγγα κτλ. Ε, η περιφερειοποίηση επίσης δεν είναι λύση. Χρησιμοποιούμε την εμπειρία των αλλήλων. Μας λένε ότι ο γάδ, ε, υπάρχει πρόβλημα με το γάζ. μα. εξηγήσουν ακριβώς τι περίπτωση πρώτη. Κυρία Λεβίν, ευχαριστούμε. Ε, μόλις είπατε αυτά που ήθελα να σχολιάσω και εγώ. Ε, είναι πολύ ευαίσθητο το περιεχόμενο, είναι υφάλμηρο το νερό και δεν μπορούν να ζήσουν πάρα πολλά είδη στη Βαλτική. Ε, και είναι συγκεκριμένη η αλυσίδα. Μιλάμε ε, για το οικοσύστημα και την προστασία του στη Βαλτική. Ε, έχει μειωθεί τόσο πολύ το απόθεμα από το 80 και μετά του γάδου που είναι κρίσιμη η κατάσταση. Και τι σημαίνει έχουμε βγάλει 60, 70 ή και 80% του ενήλικου πληθυσμού του γάδου κάθε χρόνο. Είναι πάρα πολύ πολύ αυτό και επίσης συμφωνώ με αυτό που είπατε για την υπερεκμετάλλευση της Αρδελόρεκας επί σειρά ετών. Ε, και ισχύουν αυτά που είπατε για τη Ρέγκα και τη Σαρδελόρεκα και είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά γιατί έχουν αυτή, αυτό το αποτέλεσμα ντόμινο. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση. Οι εμπειρογνώμονες ε, μας είπανε ότι λόγω της έκρηξης αρδελόρεγκας ε, δεν υπάρχει πια ζωικό πλα... που είναι η τροφή της αρδελόρεγκας. Δηλαδή η έλλειψη του ζωικού ε, πλανκτόν οδηγεί σε ευτροφισμό γιατί τα φύκια τρώνε αυτό το πλανκτόν και γι' αυτό υπάρχει ο ευτροφισμός γιατί υπάρχει μεγάλη ανισορροπία στο οικοσύστημα της Βαλτικής θεωρείται η Βαλτική ως η πλέον μολυσμένη θάλασσα. Είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η περιοχή. Είμαστε από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου και θα έπρεπε να έχουμε τους πόρους και τις έχουμε κιόλας για να προστατεύσουμε το οικοσύστημα ε, και να βρούμε ποια ε, είδη μπορούν να σωθούν σε αυτό το θαλάσσιο περιβάλλον. Ανησυχούμε για τη βιομηχανία, αλλά έχουν γίνει επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια για να, ε, για να επιστρέψουν τα αποθέματα γαδού και ρέγκας η αρχή της προφύλαξης. Ναι, συμφωνούμε. Αν δούμε ε, τους πίνακες του ISIS, ε, για, με τα διάφορα σενάρια, δηλαδή πώς πρέπει να ε, αλλιεύουμε τη Σαρδελόρεγκα και τι πρέπει να γίνει. Λέμε μείον 31% μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για την αλλιευτική δυνατότητα βάσει της αρχής της προφύλαξης. Ε, παρόλα αυτά θα μειωθεί κατά 5% το απόθεμα μέχρι το 2011. Ε, τελικά μείον 16%, μείον 25% να τα νούμερα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ούτως ή άλλως θα μειωθεί όμως η βιομάζα ανεξάρτητα τώρα από τους αστάθμιτους παράγοντες του περιβάλλοντος. Ε, ε, ε, ο ΆΙΣΕΣ προβλέπει μείωση ανάμεσα σε 10 και 15% ούτως ή άλλως. Είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου ότι για τη Βαλτική θάλασσα οφείλουμε να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύλαξης γιατί έχουμε τους πόρους, έχουμε τις γνώσεις και πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτά τα λίγα είδη που είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα και το ξέρουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Σκούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα είναι αναγκαίο επιστημονικές μελέτες να γίνουν και σίγουρα υπάρχουν μέθοδοι υπολογισμού για τη βιομάζα και πριν από αρκετά χρόνια μας είπαν ότι τα αποθέματα γάδου βρίσκονται σε τέτοια κακή κατάσταση που το καλύτερο θα ήταν απαγόρευση, απόλυτη απαγόρευση αλίευσης. Ακριβώς ε, αυτό το, η βιολογική ισορροπία που είναι αναγκαία και που έχει σχέση με μια τροφική αλυσίδα πρέπει να λαμβάνετε ιδιαίτερα υπόψη. Είναι ενδιαφέρον και αν συζητήσετε με τους ψαράδες σας, δεν ξέρω αν έχετε κάποιους τέτοιους στη Σουηδία, εμείς έχουμε ακόμα τέτοιους στην βορειοανατολική Γερμανία. Λένε αυτοί ότι τώρα εφέτος έχουμε 15% μεγαλύτερη ποσόστοση για το γάδο. Αξιοπρόσεκτο αυτό. Δόθηκαν δηλαδή ποσοστώσεις όσον αφορά υδατοκαλλιέργειες και δεν ξέρω και τι άλλο και ξαφνικά ανάκαμψε ο γάδος. Και τώρα κάθε δέκα χρόνια τι λένε οι ψαράδες. Παίρνουμε τεράστιο κύμα όθησης ε, υδάτινο που σε σχέση με το γάδο αποκαθιστά την τάξη των πραγμάτων. Κάπου πρέπει να έχουμε την πείρα που έχουν οι αλληλείς και να την λαμβάνουμε υπόψη και να τη σεβόμαστε και να μην υπολογίζουμε μόνο με μεθόδους υπολογισμού επιστημονικές αγνοώντας την πείρα των αλλιέων. Εδώ θα πρέπει να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα τι γίνεται βιολογικά και επιστημονικά με αυτό το απόθεμα. Τι γίνεται με το πλανκτόν. Τι γίνεται και τι θα γίνει με την τροφή αυτών των ψαριών στο μέλλον. Κάποια πράγματα δεν βρίσκονται σε ισορροπία. Υπάρχουν υπερβολικά προβλήματα σε σχέση με την τροφή τους. Πρέπει όλα αυτά να τα ξέρουμε πριν πει κάποιος ότι α εντάξει ωραία να περικόψουμε τα, α, τις ποσοστώσεις για τις, τα αλλιεύματα αυτά για τους αλλιείς μας. Δεν ικανοποιούμε με τέτοιες λύσεις. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά παθιασμένη αυτή η τοποθέτηση και μας εντυπωσιάζει. Δίνω τον λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Την κυρία, πώς λέγεται μια στιγμή. Γέψενα, μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για να απαντήσω στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Διαβούλευση με τους ε, Έχουμε διαβουλευτεί με τα σε τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και το ΡΑΚ της Βαλτικής ε, ενεργοποιείται ιδιαίτερος. Έχει ήδη καλές ιδέες, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και κάναμε πολύ καλή ανταλλαγή πληροφοριών. Γίνεται η διαβούλευση λοιπόν με τους αλληλείς μέσω των ΡΑΚΣ. Όταν παρουσιάσαμε τις φετινές προτάσεις για τις αλλιευτικές ε, δυνατότητες στη Βαλτική, ε, έγιναν δεκτές από το ΡΑΚ και κατανοούν την ανάγκη προστασίας του αποθέματος που είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ε, ο εργάδος ε, σε σχέση με άλλα πελαγικά είδη τώρα. Ε, ξέρετε ότι είχαμε το σχέδιο διαχείρισης του μπακαλιάρου στο, στη Βαλτική που ισχύει εδώ και χρόνια και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και έτσι φέτος μπορούμε να αυξήσουμε για το γάδο σημαντικά το τάκ. Στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου η Επιτροπή ε, συζητούσε ένα παρόμοιο πολιετές σε σχέδιο διαχείρισης για τα πελαγικά είδη για να καλύψουμε όλη την τροφική αλυσίδα, διατροφική αλυσίδα στη Βαλτική. Τουλάχιστον όλα τα είδη που έχουν κάποια εμπορική αξία. Θα καλύψουμε τη ρέγγα, τη σαρδελόρεγκα και ε, λάβαμε από τον σε επιστημονικές συμβουλές βάσει των οποίων ε, είναι σημαντικό αφού έχουμε τα ε, τελικά πορίσματα της μελέτης, θα, το ταχύτερο δυνατόν θα υποβάλουμε προτάσεις. Αυτά για το πολιετές σχέδιο διαχείρισης για τη ΡΕΚΑ και τη Σαρδελόρικα στη Βαλτική. Αυτό είναι σημαντικό για τη ρέγγα. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ε, οι κλιματικές αλλαγές, ε, για ε, τα ηχθίδια και για το γόνο και για τα αυγά, συγγνώμη, των ψαριών. Πρέπει να γίνουν μελέτες για να έχει την τεχνογνωσία ο ΆΙΣΕΣ ε, για να μας δίνει στη συνέχεια συμβουλές ε, σχετικά με αυτά τα σχέδια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούν θέλει να κάνει άλλη μια ερώτηση. Μια σύντομη επερώτηση. Μπορούμε του χρόνου το 2010 αυτό το σχέδιο διαχείρισης να το αναμένουμε, έχει προπαρασκευαστεί, είναι έτοιμο ώστε να μπορέσουμε να το εξετάσουμε και να το αντιμετωπίσουμε και να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη πολιτική για την ανάκαμψη των ρεγκών και στην ε, εκμετάλλευσή τους. Είναι ένα αίτημα αυτό, μια απέτηση από πλευράς μας να γίνει. Yes, you can for sure. Ναι, σίγουρα μπορείτε. Στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους θα είναι στη διάθεσή σας. Η κυρία Ροντούστ. Κι εγώ άλλη μια φορά μια περώτηση. Με ενδιαφέρει και είναι φλέγον αυτό. Τι γίνεται με τους γόνους της των ρεγγών. Είπατε, αρκετοί επιστήμονες λέει, ε, με, ε, κάνουν μελέτες ε, στα κράτη-μέλη, ε, συντάσσουν τις μελέτες. Ενδιαφέρον αυτό αλλά θα μου άρεσε, θα ήθελα να έχω μια συνθετική μελέτη για μας για να μπορούμε να εργαστούμε με αυτά όλα διότι δεν θα είμαστε σε θέση να πάμε στα κράτη-μέλη και να αντλήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις συλλέξουμε εμείς. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη επισκόπηση, μια τοποθέτηση από πλευρά σας. Τι γίνεται με τους γόνους των ρεγγών, διότι ακούμε από παντού ότι καταστρέφεται, δεν ανανεώνεται και χωρίς γόνους, χωρίς νέα ψάρια δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχουν ρέγγες τι θα γίνει. Γι' αυτό δεν, ξέρουμε πώ θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία εκπρόσωπο τη Επιτροπή, να απαντήσει. Uh, uh, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει παρανόηση για του χρόνου, δεν έχουμε χρήματα για ειδικέ μελέτε που αφορούν τη Ρέγκα. θα βασιστούμε για να κάνουμε το πρόγραμμα διαχείρισης στις μελέτες του ISIS και όλων των άλλων των πυρογνώμων που και όλα αυτά θα αποτελέσουν βοήθεια για μας. Βοήθημα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ καλή γιατί έχουμε χρόνο, ε. Αλλά μην νομίζετε ότι έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Κυρία Ρόντους, το λέω όμως Είμαι σήμερα πολύ ευέλικτη, δεν έχουμε χρόνο. Εν πάρτε πάλι το λόγο. Ε, όχι, δεν θέλω να διατυπώσω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ερώτηση προς την Πρόεδρό μας. Εντάξει, όταν μας λέει η Ευρωπαϊκή, μου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον προπολογισμό δεν υπάρχουν λέει κονδύλια για αυτή τη μελέτη. Εμείς όμως εδώ διαπιστώνουμε ότι πραγματικά είναι δραματική η κατάσταση όταν ο γόνος δεν μπορεί να αναπτυχθεί και να υπάρξουν νέα ψάρια και οφείλεται είτε σε αρρώστια είτε σε οποιονδήποτε άλλο λόγο. Εμείς έχουμε δυνατότητες να κάνουμε κάτι ή όχι. Δεν ξέρω αρκετά τα πράγματα, αλλά όταν γνωρίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο μείζον πρόβλημα, δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια και να πούμε δεν έχουμε κονδύλια και δεν μπορούμε να μελετήσουμε αυτό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, πώς θα γίνει, ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ πιστεύω ότι κατανόησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά που είπε. Δεν έχουμε και κονδύλιο για τέτοιου είδους ε, δράσεις, τέτοιου είδους πράγματα. Είναι ένα πράγμα που δεν είναι ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Εγώ κατανόησα από όσα είπε εκπρόσωπος Επιτροπής ότι χρησιμοποιούν, λέει, τα μέσα τα κανονικά που έχουν για οποιαδήποτε αποτίμηση αποθεμάτων. Το όργανο που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αποθεμάτων από τις Ρέγγες μέχρι οποιοδήποτε άλλο. Εδώ είναι η ίσες που κάνει την ετήσια αξιολόγηση, αποτίμηση των αποθεμάτων και λέει αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει η Ρέγγα της Φαλτικής για παράδειγμα και με αυτά τα χαρακτηριστικά και τις συστάσεις ε, που η ίσες ε, διατυπώνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπιπλέον και υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση δεν το ξέρω, αλλά για την, ε, ε, για την ε, αντσούγα για παράδειγμα, τη σαρδέλα υπάρχουν μέσα όργανα, έχουμε και το Ισπανικό Ίδρυμα που εργάζεται και συνεργάζεται και είναι αυτό το οποίο είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για τη Βαλτική εδώ. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία υπάρχουν δυνατότητες για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να αυξηθούν αυτά τα κονδύλια, αυτά τα μέσα, αλλά υπάρχει αξιολόγηση που γίνεται για κάθε ένα από τα αποθέματα ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω αν θα, ήθελε, θα θέλατε περισσότερο να εμβαθύνετε σε κάποιο τέτοιο θέμα, αλλά η αξιολόγηση γίνεται ω ήθιστε για κάποια είδη και εδώ γίνεται λόγος και για κάποια άλλες φορές πελαγικά είδη, άλλες φορές κάποια κυκλικά ανακυκλούμενα στην εξέλιξή τους είδη και υπάρχουν μια σειρά παράγοντες που δεν είναι πάντα εύκολο να αξιολογηθούν, να αποτιμηθούν για παράδειγμα σε σχέση με, τις, ε, με, με είδη θαλάσσια που λόγω της βιολογικής τους ε, ας το πω έτσι εξέλιξης είναι πιο εύκολα. Τα πελαγικά είδη είναι πιο κυκλικού χαρακτήρα και μπορούν να υπάρξουν εδώ επιρροή ή να υπάρξει επιρροή και των ε, κλιματικών αλλαγών. Άλλες φορές πρέπει εδώ να δούμε κάποια άλλα στοιχεία, υπάρχουν και αβεβαιότητες. Παρ' αυτά Υπάρχουν ήδη που είναι πιο περίπλοκα. Εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη και επαίων με αυτά τα θέματα. Αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω είναι αρκετά σωστό. Κάθε έτος γίνονται οι αναγκαίε αποτιμήσει και αξιολογήσει. Θα γίνουν αυτά. Τα εθνικά ιδρύματα που εμπλέκονται θα δράσουν ε, είναι τα ιδρύματα των κρατών μελών που παράδειγμα, για παράδειγμα ψαρεύουν στη Βαλτική θάλασσα Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη σας ερώτηση, εμείς αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ε, να ζητήσουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη της επιστημονικής δράσης, μεγαλύτερη πρικοδότηση με κονδύλια τέτοιου είδους ε, ε, δράσεων, ώστε από πλευρά του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ανταποκριθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα πολύ περισσότερο. Θα δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να προσθέσει κάτι σε σχέση με το αίτημα της κυρίας Ρόντους. Παρακαλώ. No, indeed, madam, I, I really... Όχι, κυρία Πρόεδρε, πραγματικά δεν έχω τίποτε περισσότερο να προσθέσω μετά από αυτά τα οποία είπατε. Εξηγήσατε πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση και πώς επιστημονική αρρωγή παρέχεται από την πείρα των διαφόρων Ινστιτούτων, οργανισμών που έχουν τις γνώσεις, τις επιστημονικές, κάνουν τις μελέτες οι πραγματογνώμονες τους συνδυάζουν στα πλαίσια του ISIS. και συνεισφέρουν ο καθένας με την δική του εθνική εμπειρία ώστε να έχουμε όλα τα στοιχεία αυτά σε επίπεδο ISIS. Το εξηγήσατε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καμιά άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω να υπάρχει. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Επιτροπής και όλους τους παρεμβαίνοντες. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση του σημείου 15 και περνούμε στο επόμενο, το 16. Ανταλλαγή απόψεων για τις αλληλευτικές δυνατότητες στη Μαύρη Θάλασσα το 2010. Η Κομισιόν θα μας εξηγήσει κάποια θέματα και ο κύριος Μαρινέσκου που είναι παρόν θέλει να ζητήσει κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις. Πρώτα στον κύριο Μαρινέσκου δίνω το λόγο και μετά στην Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε στη μερίσια διάταξη το θέμα αυτό. Όπως γνωρίζετε, υπέβαλε πρόταση η Επιτροπή για κανονισμό του Συμβουλίου για τα θέματα που αφορούν ποσοστώσεις αλλιευμάτων το 2010 στην Μαύρη Θάλασσα. Εδώ προτείνεται μείωση του ΤΑΚ για την Ρουμανία και την Βουλγαρία από 100 τόνους 63 τόνους στο γύρο, βάσει συστάσεων που έκαναν εμπειρογνώμονες από την Επιστημονική Γνωγική Επιτροπή. Στην πρόταση αυτή δεν περιλαμβάνεται η ρήτρα αναθεώρησης, ώστε ενδεχομένως τον μεθεπόμενο χρόνο να επανέλθουν βάσει επιστημονικών στοιχείων τα επίπεδα των ΤΑΚ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατανοώ πάρα πολύ καλά Ποια ήταν τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Επιτροπή αυτή, η Ειδική Επιτροπή, για να υποβάλει αυτή την σύσταση. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι μέλος της υποομάδας της Μαύρης Θάλασσας, όπου δεν έγινε ποτέ αναφορά στη μείωση των ποσοστώσεων. Αποτελέσματα των μελέτων που έγιναν από τους εμπειρογνώμονες, τους Ρουμανούς και τους Βουλγαρούς βλέπουν ότι υπάρχουν αύξηση των αποθεμάτων και αυτό θα ισχύσει και του χρόνου. Εμείς είμαστε σίγουροι βάσει των στοιχείων ότι δεν έχουν τα ανώτατα επιτρεπόμενα ε, αλλιεύματα. Και πήραμε και μέτρα ώστε να μπορέσουμε τα διάφορα αποθέματα να τα ανανεώσουμε και να μειωθούν και οι διάφορες αλληλευτικές προσπάθειες. Μετά την ε, απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Όσον αφορά την ύλη του Σνάκα. επεκτείναμε στις εκβολές του Δούναμι, στις εκβολές του Δούναμι την ε, αλληλευτική μας ε, ζώνη. Plan. Ε, so, following this, Μετά, μάλλον, Μετά από όλα αυτά, η Επιτροπή Οικονομική, Τεχνητή Επιστημονική Επιτροπή πρότεινε να μειωθούν στα ποσοστά που προανέφερα τα ανώτατα επιτρεπτά λιεύματα. Μειώθηκε λοιπόν μείωση του κατά 24% για το 2001. Εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε το 2010 και να μπορέσει ό,τι γίνει να γίνει βάση ενός μηχανισμού διαφανούς ώστε να μπορούν όλες οι επιστημονικές, όλα τα επιστημονικά ευρήματα να χρησιμοποιούνται με τον ίδιο ορθολογιστικό τρόπο. Υπάρχει έτοιμο εκ μέρους μας να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί με την ε, διαχείριση όλων των άλλων, πάντως να πρέσει τις μαύρες θάλασσα και στον οργανισμό αυτόν συμπεριληφθούν όλες οι χώρες που βρέχει η μαύρη θάλασσα. Προτείνω λοιπόν πυρογνώμονες, ε, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες να, και πυρογνώμονες από την Κομισιό επίσης να δουν όλα αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Ο κύριος Μαλέκ μέρους της ε, Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος πώς μπορεί να δώσει κάποια απάντηση σε αυτό το θέμα η Επιτροπή, διότι, όπως ξέρετε, έγινε αναφορά στις ναι, κανονισμό που αφορά τα ΤΑΚ. Και αναφέρθηκε εδώ ο κανονισμός συμβουλίου. Τι ρόλο έχουμε να παίξουμε εμείς ως Κομισιόν. Από ό,τι καταλάβαμε, εμείς θα γινόταν γενικά μία ανταλλαγή απόψεων για την διαχείριση των αλλιευμάτων στη Μαύρη Θάλασσα. Πράγμα το οποίο βεβαίως όλες τις χώρες της περιοχής την αφορούν. Αλλά έχω μπλέξει εδώ. Εμεί εκ μέρου του Συμβουλίου δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εμεί είμαστε η Επιτροπή. Κύριε Μαρινέσκου, θέλετε να κάνετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση στην Κομισιά και να υποφεληθείτε από την παρουσία της. Διαφορετικά λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία είπατε, αλλά αν δεν έχετε κάτι συγκεκριμένο να ερωτήσετε την Κομισιόν, δεν είναι παρόν το Συμβούλιο για να απαντήσει. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση, διότι δεν καταλαβαίνω γιατί τον Απρίλιο η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αύξηση των ποσοστώσεων, των τάξ, κατά 25% βάσει προτάσεων που υπέβαλε η υποομάδα και η απόφαση εκ των υστέρων ήταν όχι μόνο να διατηρηθεί το παρόν επίπεδο, ούτε να αυξηθεί, αλλά να μειωθεί. Και αυτή η πρόταση συμπεριλήφθη στην πρόταση που υπευλήφθη για κανονισμό του Συμβουλίου. Θα ήθελα και πάλι να υποβάλω το εξωτερικό στην Επιτροπή. Ποια είναι τα δεδομένα που χρησιμοποιεί όταν για να λάβει τέτοιου είδου αποφάσεις. Τα δεδομένα της υποομάδας συμπεριλαμβανομένων και των εμπειρογνωμόνων από τις χώρες που βρέχουν τη Μαύρη Θάλασσα ή τα δεδομένα της Επιτροπής που δεν συμπεριλαμβάνει εμπειρογνώμονες από τις χώρες αυτές. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι μπερδεμένο είμαι για αυτή την απόφαση. Από δύο μπερδεμένε λοιπόν και συγκεχημένε καταστάσεις ίσω μπορούμε να καταλήξουμε σε μια σαφή απάντηση. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ίσως θα πρέπει να καθορίσω το εξής. Δεν με μπερδεύει η διαδικασία βάσει της οποίας η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για κανονισμό των ποσοστώσεων, το tax στην Μαύρη Θάλασσα, όπως έκανε το 2008-2009 αυτό που με απασχολεί είναι γιατί στην Επιτροπή Αλληλείας του Κοινοβουλίου μου κάνετε ερωτήσεις που αφορούν ένα κανονισμό που βρίσκεται υπό εξεργασία του Συμβούλιο. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο συνήθως. Τώρα, όσον αφορά το, ερώτησα, ερώτημα της επιστημονικής διαδικασίας που ακολουθείτε, είναι η ίδια με αυτή που ακολουθείτε και για τις άλλες ε, ε, περιοχές. Δηλαδή έχουμε την επιστημονική αισθησίας επιτροπή που πρώτα απ' όλα τεντράζει για θέματα Μεσογείου, μαύρη θάλασσα και έχουμε εμπειρογνώμονες και από τις χώρες που είναι κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, Ουλή, την Ουκρανία, την Τουρκία που συμμετέχουν στην υποομάδα συλλέγουν, αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία στην ε, ολομέλεια της CTCF υποβάλλουν τα στοιχεία και η CTCF γνωμοδοτεί. Έτσι γίνεται όχι μόνο για αυτή την αλληλευτική περιοχή, αλλά και για όλε τι άλλε συμπεριλαμβάνει και τη Βαλτική που μόλι τώρα συζητήσαμε. Δεν υπάρχει λοιπόν στην προσέγγιση καμία διαφορά. Όσον αφορά το θέμα τη σύσταση Ενό διεθνούς πολυμερούς οργανισμού για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Ήδη εξηγήσαμε και στους Ρωμάνους και στους Βουλγαρούς και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο επίσης ε, έχει συζητηθεί και εδώ, ότι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή για τη Μαύρη Θάλασσα είναι ότι η σύμβαση του Βουκουρεστίου Τροπή Μαύρης Θάλασσας που αυτή τη στιγμή έχουν εντολή για θέματα περιβαλλοντικά, μπορούν ενδεχομένως να δουν να επεκτείνεται η εντολή τους για θέματα αλληλείας στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά όλα τα μέλη της οργάνωσης αυτής δεν θα ήθελαν να αποτελέσει αυτή την οργάνωση πληρεσμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, προς το παρόν, πρέπει να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της που ασχολείται με τα θέματα της περιοχής ε, της Μεσογείου που είναι εκεί κοντά και να ακολουθείτε και για τη Μαύρη Θάλασσα η ίδια διαδικασία. Και η Ρουμανική Βουλγαρία και η Τουρκία είναι μέλη της GFCM. Ήδη λοιπόν υπάρχει ένα βήμα, ένας χώρος στον οποίο τέτοιου συζητήσεις μπορεί να γίνουν. Σας ευχαριστώ κύριε Μαλέτ. Άρα ολοκληρώθηκε το θέμα. Αυτό ήθελε ο κ. Μαρινέσκου να προσθέσει κάτι άλλο. Ναι, νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι πρόκειτο για απάντηση, διότι η ερώτησή μου κυρίως είναι για ποιο λόγο η Επιτροπή έλαβε υπόψη την πρόταση της κομίτη, της άλλης επιτροπής και όχι της υποομάδας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ειδικοί επί αυτού του θέματος και από την επιτροπή. Και η Τίδη ζήτησε η ποσόστοση του 2010 να είναι παραφερής η ίδια με αυτή του 2009. Η απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής ελήφθη και προτάθηκε η μείωση των ποσοστώσεων. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Γιατί λοιπόν έχουμε μία επιστημονική υποδομάδα αν δεν λαμβάνουμε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της. Ακούστε, εγώ δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι ρωτάτε. Κύριε Μαλέτ, θέλετε να απαντήσετε. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ καλά τίποτα. Αν είστε όμως πιο ευφύς κύριε Μάλετ, μπορεί και να την καταλάβετε εσείς και να απαντήσετε. Um, I, πρόεδρε. Δεν μπορώ να απαντήσω μια ερώτηση. Πιο πολύ από ό,τι έκανα. Εγώ διε, περιέγραψα τη διαδικασία και είπα ότι η διαδικασία είναι η ίδια με αυτή την οποία ακολουθούμε στα πλαίσια αυτών των επιτροπών και υποομάδων με τη συλλογή και αντιπαραβολή στοιχείων που κάνουν και όλες τις άλλες αλληλευτικές περιοχές. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα άλλο. Και όπως σας είπα, από θεσμικής πλευράς είναι λίγο αυτό που συζητείτε εδώ. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εξετάζει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο και θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Ελίας τον Νοέμβριο. Είναι λοιπόν κάπως λεπτά τα πράγματα. Εντάξει, θα περιμένουμε λοιπόν να γίνει το Συμβούλιο Αλληγίας τον Νοέμβριο. Κύριε Μαρινέσκου, θα δείτε σε ποιον ε, θα υποβάλλετε κριτικές και αν θα ζητήσετε εξηγήσει. Ευχαριστώ κύριε Μαλέτ. Άρα το σημείο 16 ολοκληρώθηκε. Περνάμε στο επόμενο. 17. Αλία στην περιοχή της Συμφωνίας της ΓΙΑΜ. Γενική Επιτροπή Αλλιέ για τη Μεσόγειο. Ο κύριος Ριμπελίνη είναι ο εισηγητής. Δεν είναι εδώ σήμερα ο κύριος Ριμπελίνη. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν μεταφορά στι εθνικέ μα. Μου λένε ότι η Επιτροπή δεν έχει κανένα πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο ορίσει η Επιτροπή μα. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Ανταλλαγή απόψεων 4 Νοεμβρίου, παρουσίαση του σχεδίου έκθεση 30, ψηφοφορία στην Επιτροπή 27-28 Ιανουαρίου 2010. και στην πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου ψηφοφορία. Μου λέτε ότι η Κομισιόν δεν έχει με το χρονοδιάγραμμα πρόγραμμα. Άρα θα ενεργήσουμε ως εξή. Λοιπόν, 18. Τα διάφορα. Θέλει κανένα συνάδελφο κάποιο πρόβλημα να θέσει. Εάν όχι, το επόμενο. Ανακοίνωση Πρόεδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν οι συντονιστέ. διανεμήθηκε σήμερα το έγγραφο που αφορά τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές στη συνεδρίαση πες το απόγευμα. Σας τις υποβάλλω. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε πολύ καλοί. Λίγοι, αλλά καλοί. Και πρέπει να σας πω ότι το κείμενο του ήταν της ερώτησης, η σας απεστάλλει χθες, έχει προθεσμία ως την Παρασκευή το μεσημέρι για να υποβάλλετε παρατηρήσεις, εάν έχετε να υποβάλλετε παρατηρήσεις. Διαφορετικά θα θεωρήσουμε το κείμενο μπορεί να αποσταλεί ως έχει τη διάσκεψη των πρόεδρων. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίθησαν οι αποφάσεις, περίπου στο τελευταίο σημείο, η ημερομηνία της προσεχούς συνεδρίασης, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες από τις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους διαρμηνείς. Λύε τη συνεδρίαση.